Ευχαριστώ. Αλλά καθίστε. Γιατί έχουμε εδώ μιλητή. Μπορεί να μην έχουν έρθει πολλοί βουλευτέ, αλλά εμείς πάντως θα τα κάνουμε όλα κανονικά αν βγει κανείς μπορεί και να τα διαδώσετε ότι έχουμε οργανώσει αυτή τη συνάντηση και να έρθουν. Λοιπόν, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχει καμία αντίρρηση. Όχι. Ε, τότε εγκρίνεται. Έχουμε και Charles κουτ Και για σήμερα και για αύριο. Θα αλλάξει βέβαια, άλλη σήμερα, άλλη αύριο. Έχουμε και ένα νέο μέλος, την Άννη Ποδηματά, που θα αντικαταστήσει τον Ιτίν Ντανιέλης. Και τώρα το σημείο 3. Ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Ιωβανίνη Καρόσιο είναι η πρώτη του εμφάνιση στην Επιτροπή μας εικόν της οποίας μία από τα καθήκοντα είναι να είναι ένα ελέγχει τις δραστηριότητες της λεγόμενης Επιτροπής Λαμφαλούς 2. Και αυτό το κάνει με μια παρουσίαση 15 λεπτή περίπου και μετά γύρω ερωταπανδύσεων. Η δε εισήγηση θα είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα. To So Σας συγχαίρω λοιπόν για τον διορισμό σας και σας καλωσορίζω εδώ στην πρώτη επίσκεψη της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Με μεγάλη χαρά και αίσθημα τιμής προσήλθα εδώ σήμερα για να συνεχίσουμε το διάλογο που είχατε αρχίσει με τον προκάτοχό μου. Οι αποφάσεις της Επιτροπής σας και οι απόψεις σας είναι ουσιώδης για μας. Η οργάνωσή μας, η ΕΕΑΤ, όπως ξέρετε, είναι πολύ σημαντική για να ελέγχει τις εποπτικές ε, διαδικασίες των τραπεζών και για να πραγματοποιεί μια ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών μεταξύ των μελών της. Στην αρχή στοχεύαμε μόνο τους στόχους της Βασιλείας 2 και σε αυτή τη βάση γράφτηκαν πολλές κατευθυντήριες γραμμές και καθώς και με βάση την οδηγία που μετέφρασε τη Βασιλεία 2 σε ευρωπαϊκούς όρους. Μετά όμως διευρύναμε το, την εντολή μας και στην ανάλυση των κινδύνων. Ο συντονισμός των εποπτικών δραστηριοτήτων επίσης δεν παρέμεινε ουσιώδης ως κέντρο ενός δικτύου Ευρωπαίων εποπτών. Επίσης, τη αιτήση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών μπορούμε να απαντούμε σε ερωτήματα και απορίες όπως ε, τι, τι μέτρα πρέπει να λαμβάνονται όταν δεν υπάρχει ρευστότης, όταν σημειώνεται ή ξεσπάει κρίση κτλ. Σήμερα θα βασιστώ σε τρία κυρίω θέματα. Τη νέα ευρωπαϊκή δημοσιονομική αρχιτεκτονική, τη δέσμη προτάσεων της Επιτροπής της Βασιλείας για την Εποπτεία των Τραπεζών και τις προτεραιότητες μας για το 2010. Για την αρχιτεκτονική, δημοσιονομική αρχιτεκτονική, εμείς στηρίζουμε τα αποτελέσματα της έκθεσης Ντελαροζιέρα και της προτάσεις της Επιτροπής στην οποία βασίζεται. Η πολιτική συζήτηση οδήγησε σε σημαντικές αναπροσαρμογές ε, και η δέσμη μέτρο προέβλεπε το Συμβούλιο να χορηγεί στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή τα εργαλεία και τις ευθύνες που χρειάζεται πράγμα το οποίο είναι μεγάλη πρόοδος σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. Το πιο ζωτικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής αυτής είναι ότι επιτρέπει στις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές να εφαρμόζουν γνωστά και διεθνή πρότυπα που να είναι εφαρμόσιμα σε όλες τις χώρες μέλη χωρίς να χρειάζεται εθνική έγκριση χωριστά. Και αυτό για να υπάρχει μεγαλύτερη συνέπεια στην εφαρμογή των δημοσιονομικών μέτρων. Και εμείς δεχόμαστε τα μέτρα αυτά και την δημιουργία ενιαίου συστήματος τραπεζικών κανόνων που θα εμφαίνονται στην οδηγία Omnibus. Η εντολή προβλέπεται να καλύπτει όλους τους κύριους τομείς της διευθέτησης των τραπεζικών σύμφωνα με τις προτάσεις του Συμβουλίου Δημοσιονομικής Σταθερότητας και των τελευταίων αποφάσεων του ΓΑΜΑ 20. Θέλουμε επίσης τις αλλαγές αυτές να τις συμπεριλάβουμε στη Γενική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία με τρόπο ώστε να είναι σίγουρη και βέβαιη η εναρμονισμένη εφαρμογή των κανόνων. Αυτό βέβαια ελπίζουμε να καταλήξει σε μεγαλύτερη προστασία των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη ε, ως προς το κόστος που θα έχει οποιαδήποτε δημοσιονομική διαμεσολάβηση για να διασφαλιστεί έτσι απρόσκοπτη ανάπτυξη. Λόγω της τεχνογνωσίας που έχουν οι επόπτες θα πρέπει να έχουν τον κύριο λόγο κατά τον καθορισμό των μελλοντικών πανενοσιακών προτύπων, τεχνικών προτύπων. Και η έγκριση τους από την Κομισιόν πρέπει να περιοριστεί σε μια απλή αναθεώρηση μετά από την έγκριση των προτύπων που θα συγγράψουν οι επόπτες, η, ανα... η έγκρισή τους από την Κομισιόν πρέπει να περιοριστεί σε μια αναθεώρηση του νομοτύπου ή μη των εφόσον βέβαια και, η Ευρωπα... και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο συμφωνεί. Δηλαδή πιστεύουμε ότι η έγκριση της Κομισιόν δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα μετατροπής των προτύπων αυτών. Αυτό θέλουμε να λέγεται ρητά στις τελευταίες γραμμές του σχετικού κανονισμού ή απόφασης. Θα δημιουργηθούν κολέγια εποπτικά τα οποία με τη σειρά της θα επιβλέπει η οργάνωσή μας πανενοσιακός. Υπάρχει κολέγιο εποπτών για 35 μεγάλους τραπεζικούς ομίλους και το 2010 θα καθορίσουμε και καινούριου στόχους για καθορισμό νέων εποπτικών κολεγίων και για άλλους τραπεζικούς ομίλους. Πέρα από αυτά τα κολέγια που υπάρχουν θα καθορίσουμε στόχους και για να μπορούν αυτά να κάνουν συνδυασμένου ανάλυση του κινδύνου υπό τους κανόνες του πυλώνα 2. Είναι ζωτικό η δημοσιονομική αυτή αρχιτεκτονική να διευκολύνει την εργασία των κολεγίων αυτών. Οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ κολεγίων και εποπτών θα διευκολύνονται καθώς και μεταξύ μεγάλων ε, δημοσιονομικών ομίλων και εποπτών. Θα γίνονται περιοδικές αναθεωρήσεις ή αξιολογήσεις μαζί με τις αναλύσεις που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, Ανάλυσης Συστημικών Κινδύνων έτσι ώστε να υπάρξει μια ταύτιση των ε, κινδύνων που μπορούν να, να αφήσουν ή να ξεσπάσουν, πράγμα το οποίο εμερικώς κάνει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά τα κολέγια των εποπτών θα κάνουν δική τους αξιολόγηση και τις επιπτώσεις που προβλέπουν σε μεμονωμένους ομίλους. Η οργάνωσή μας, η ΕΑΤ, είχε αρχίσει ήδη και πέρυσι να προσχεδιάζει αυτή τη δραστηριότητα και το 2010 θα συνεχιστεί σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναγνωρίζουμε επίσης την ανάγκη που υπάρχει να γίνουν γνωστά περισσότερα στοιχεία ανατομέα λόγω της ίδιας της φύσης του δημοσιονομικού κινδύνου που μπορεί να προκύψει. Παρ' όλα αυτά, η κρίση μας έδειξε ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα στοιχεία ανατομέα. Γι' αυτό έχουμε πολύ μεγαλύτερη συνεργασία με τους ανάλογους οργανισμούς και γι' αυτό τονίζουμε πόσο σημαντική είναι η συνεργασία αυτή στη νέα αρχιτεκτονική. Διότι έτσι θα μπορέσουμε να ταυτίσουμε ποιοι είναι όντως οι κοινοί κίνδυνοι σε θέματα όπου επικαλύπτονται πολλοί τομείς. Αυτό ήταν το πρώτο θέμα. Τώρα το δεύτερο. Οι νέες προτάσεις αναθεώρησης των τραπεζικών κανονισμών. Η οποιαδήποτε λύση και να δοθεί πρέπει να είναι σφαιρική. Το 9 η Επιτροπή της Βασιλείας ακολούθησε τις, τα συμπεράσματα του ΓΑΜΑ 20 και οι προτάσεις της θα διατυπωθούν φέτος και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από το 12. Προβλέπονται βελτιώσεις στην ε, ασφάλιση των παρακινδυνευμένων κεφαλαίων, ιδίως σε περιπτώσεις κρίσης, μέτρα αντιμετώπισης κυκλικών κρίσεων και οι επιπτώσεις όλων όλης αυτής της νομοθεσίας θα φανούν από μία μελέτη με χωριστή. Και το δείγμα που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι διευρυμένο σε σχέση με προηγούμενες όπου, ε, μελέτες όπως και πιο μικρομεσαία τραπεζικά ιδρύματα. Επίσης, θα μπορέσουμε να δούμε τι επιπτώσεις έχουν οι εναλλακτικοί ορισμοί που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Ένωσης. Τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο θα φανούν όλα αυτά. Θα θέλαμε επίσης να δοθούν θετικά κίνητρα σε ορισμένους τύπους επιχειρήσεων που θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνες σε περίπτωση δημοσιονομικής κρίσης. παραδείγματο χάρη μεταξύ, ε, μέσω ρητρών που να επιτρέπουν τη χορήγηση υψηλών ποσών. Έχει ζητηθεί επίσης από την οργάνωσή μας να προταθούν μέτρα για ιδιαίτερα προβληματικούς τομείς, αλλά θα περιοριστώ σε ένα. Αξιολόγηση των μίνιμουμ απαιτήσεων για κατακράτηση κεφαλαίων. Κάτι το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους επενδυτές, αλλά δεν είναι ούτε αυτό καμία πανάκια, ακόμη και σε περίπτωση κρίσης. Και θα προτιμώνται άλλα μέτρα. Εμείς πιστεύουμε ότι όλες οι εναλλακτικές λύσεις κατακράτησης που προτείνονται μπορούν να κρατηθούν αλλά μόνο μέχρι 5% διότι μεγαλύτερη αύξηση θα μπορούσε να υπονομεύσει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν κρίσεις. Και στα Ηνωμένα Πολιτείας κάτι ανάλογο έχει προβλεφθεί. ώστε να διευκολύνεται η χορήγηση καλύτερης ποιότητας δανείων. Για τα έσοδα των τραπεζών, με βάση πάντα τις προτάσεις της Βασιλείας, θα καθορίσουμε ορισμένα πρότυπα που πρέπει να ακολουθούν οι τράπεζες για να μην ενθαρρύνουν την ανάληψη υπερβολικού κινδύνου. Τώρα έχουμε τη δικαιοδοσία να καθορίσουμε κατευθυντήριες γραμμές για να μπορούμε να βοηθήσουμε εταιρείε σε περίπτωση κρίσης, πράγμα το οποίο θα γίνεται σε δύο φάσεις, θα γίνει σε δύο φάσεις, μια μία-μία μελέτη σε δύο φάσεις. Πρώτον, να δούμε πώς εφαρμόστηκαν σε εθνικές περιπτώσεις τα κριτήρια αυτά και δεύτερον πώς αντέδρασαν τα χρηματοπιστωτικά ιδουρήματα. Τέλος, ποιες είναι οι προτεραιότητες της ΕΑΤ για το 2010. Η υψηλότερη θα είναι καλύτερη εποπτεία και αντιμετώπιση της κρίσης. Οι προβλεπόμενες αλλαγές στη Βασιλεία 2 και επίσης η προβλεπόμενη μεταφορά δικαιοδοσιών από την ΕΑΤΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τέλος πάντων στην ΕΜΠΑ όπως λέμε, και θα καθορίσουμε και γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο λειτουργίας των εποπτικών κολεγίων και τη γενικότερη διαχείριση του κινδύνου πέρα από όσα είχαμε ήδη αναλάχεις να αναλαμβάνουμε το 2009. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την αποκάλυψη στοιχείων επίσης, disclosure δηλαδή, έχουν ήδη αναλυθεί σε πρώτη φάση για ορισμένες τράπεζες που θα αναγκαστούν να συμμορφωθούν με τις γραμμές του, της ΕΑΤ. Επίσης, έχουμε συμβάλει στην εργασία της Κομισιόν για τη δημιουργία ενός γενικότερου πλαισίου διατραπεζικής διαχείρισης του κινδύνου. Και το πλαίσιο αυτό στοχεύει όλοι οι εθνικοί επόπτες στην Ένωση να έχουν επαρκή και κοινά εργαλεία για να μπορούν να ταυτίσουν εγκαίρως προβλήματα και να μπορούν να παρεμβαίνουν ώστε τα προβλήματα αυτά να επιλύνονται ακόμη και στην περίπτωση που ορισμένες θηγατρικές τραπεζών έχουν, ε, ανήκουν σε διαφορετικές εποπτικές δικαιοδοσίες από την μητρική. Επίσης έχουμε ταυτίσει και άλλα μια σειρά μέτρων για παρεμβάσεις, εργαλειοθήκη ολόκληρη για κάθε χώρα μέλος. Έπειτα πρέπει να ε, πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες για να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία αυτά επειδή θα έχουν επιπτώσεις στα κέρδη των μετόχων. Θα υπάρχουν ορισμένα συγκεκριμένα κριτήρια και όχι αυτόματα. Χρειάζεται βέβαια για να εφαρμοστεί αυτό ενισχυμένο πλαίσιο συνεργασίας ή πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας. Γιατί θα μπορεί να, μπορεί να χρειαστούν κοινά μέτρα από κοινού περισσότερες από μία χώρες. Οι εγγυήσει θα συμβάλλουν και αυτές με τα υπόλοιπα μέτρα. Θα υπήρχε όμως και η λύση της δημιουργίας μεγαλύτερης αλληλεγγύης μέσω ενός αμοιβαίου μηχανισμού εγγυήσεων και ασφάλειας όποτε χρειάζεται. Τέλος, για τις πιτοχεύσεις οι τροποποιήσεις του σχετικού νόμου που αφορούν διαμεθοριακές τράπεζες θα τροποποιηθούν και η νέα αυτή δομή πρέπει, η δομή πρέπει να τύχει συντονισμού με τις δικαιοδοσίες που θα χορηγηθούν στην λεγόμενη ΕΜΠΑ. ΕΜΠΑ. Thank σας κατευχαριστώ. Κοιτάξτε, θα καταλάβατε ότι κάνα δυο κομμάτια τα πήδηξε ο μιλητής γιατί βιαζότανε, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Muchas gracias, señor presidente. Estamos aquí. βρισκόμαστε οι δύο εισηγητές, ο κύριος Βίγκο και εγώ, σε σχέση με τον Οργανισμό Τραπεζικής Εποπτείας. Και βεβαίως θα πρέπει ο κύριος Βίγκο να μιλήσει και εξ ονόματος Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, ενώ εγώ θα προωθήσω την άποψη της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής. Το θέμα των ε, τεχνικών προδιαγραφών επιλύεται αν θεωρήσουμε ότι πρόκειται για ε, πράξεις πληρεξουσιότητας εδώ και η Επιτροπή είναι εκείνη η οποία θα εγκρίνει τις προτάσεις της ε, Εποπτικής Αρχής. Ως προς τις διασυνοριακές αρχές, όπως ε, αναφέραμε με, τον, ε, με την κυρία Φερέιρα, έχουν ως εξής. Από το 2000, από τότε που άρχισε να λειτουργεί η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Υποθέσεων, εμείς ε, ταχθήκαμε υπέρ του γεγονότος ότι η απελευθέρωση των αγορών σημαίνει ότι οι χρηματοπιστωτικοί φορείς μπορούν να δράσουν απρόσκοπτα, ενώ το θέμα της εποπτείας έλυγε στα εθνικά σύνορα. Άρα προωθήσαμε μια γενικότερη εποπτεία, η οποία όμως δεν λειτουργήσε και μετά ανέκυψε και η κρίση. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μία πραγματική ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτική αρχή η οποία να ασχολείται με ε, διασυνοριακά ζητήματα συστηματικού κινδύνου και με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να δράσουμε χωρίς να, να δημιουργήσουμε περαιτέρω γραφειοκρατία με βάση τις ε, εθνικές τραπεζικές αρχές εποπτείας που θα ήταν εξουσιοδοτημένοι φορείς και θα λειτουργούσαν με βάση τις ε, εποπτικές εντολές του Ευρωπαϊκού Διατραπεζικού Φορέα. Τώρα το ζήτημα είναι ποιος θα καταβάλει τα έξοδα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να, δημιουργήσει, να δημιουργηθεί ένα ειδικό ταμείο ή ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο θα ήταν υποχρεωμένο έτσι ε, ώστε να εγγυηθεί για τις καταθέσεις για να μην τεθεί σε κίνδυνο το σύστημα. Εάν αυτά τα κονδύλια είναι ανεπαρκή, όπως σε περίπτωση κρίσης, θα μπορούσαμε να προβούμε σε περαιτέρω ε, σε μια περαιτέρω δράση η οποία θα βαζιζόταν και σε έκδοση ομολογιών. Αν παρίστατο ανάγκη υπάρχουν νομικά και θεσμικά ζητήματα, αλλά εδώ πρόκειται για μια πρώτη σκέψη, πρώτη συλλογιστική. Θα πρέπει, θα ήταν συνετό να έχουμε μια ευρωπαϊκή εποπτική αρχή για τους ε, συστηματικούς κινδύνους ή συστημικούς κινδύνους που γνωρίζει το σύστημα με βάση ένα ταμείο το οποίο θα χρηματοδοτήσει αυτή τη δραστηριότητα έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ε, καταβολής του αντιτίμου από τους καταναλωτές, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για καταθέσεις για τις οποίες κάποιος θα πρέπει να εγγυηθεί σε περίπτωση κρίσης. Απάντηση. Θα ξεκινήσω το τέλος το ερώτημα του ποιο θα πληρώσει σε περίπτωση κρίσης διασυνοριακών ε, ε, τραπεζών. Είναι κρίσιμο το ερώτημα αυτό και για τη διάρκεια της κρίσης της δημοσιονομικής ε, το είδαμε. Ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους η λύση που βρήκαμε τελικά, μάλλον δεν ήταν και η καλύτερη. Σε πολλές περιπτώσεις Είχαμε διαφορετική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της κρίσης στους διάφορους συνοριακούς ε, φορείς. Θα μπορούσαμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό έχοντας κάποιες συμφωνίες μεταξύ των εποπτικών αρχών, των ελεγκτών που ελέγχουν μία συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο όμιλο και αυτές οι συμφωνίες ήδη συνάπτονται στα πλαίσια του κολεγίου Τη δουλειά που, που κάνουν τα κολέγια. Αυτέ οι συμφωνίε θα μπορούσαν να επεκταθούν ώστε να καλύπτουν και την παρέμβαση και την επίλυση των κρίσεων. Θα ακούσατε ήδη ότι προτείνονται νέοι τρόποι για την αντιμετώπιση των τέτοιου είδους προβλημάτων έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε κατά πόσο κάποιες ομάδες που μπορεί να είναι ε, πιο ευάλωτες ε, από συστημικής πλευράς ε, πρέπει να αντιμετωπιστούν με καλύτερα μέτρα. Πώς μπορούμε λοιπόν να συνδυάσουμε όλα αυτά τα στοιχεία και σε επίπεδο διασυνοριακό. Αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί για να καλύψει και το θέμα αυτό. Το πώς δηλαδή όλα αυτά τα, όλες αυτές οι εταιρείες από ενός ομίλου θα μπορέσουν να σωθούν σε περίπτωση κρίσης και ποιος θα καταβάλει τα έξοδα. Η εκ των προτέρων ε, ε, παρέμβαση που θα πρέπει να γίνει στην περίπτωση αυτή θα γίνει για να εξασφαλίσουμε ότι οι ελεγκτές, οι επόπτες συμφωνούν με τη δομή του ομίλου, της, ε, του τραπεζικού ομίλου και θεωρούν ότι είναι ασφαλέ, ασφαλής ώστε ακόμη και σε περίπτωση ε, κρίσης να μπορέσει να είναι αποδοτικός, αποτελεσματικός. Τώρα, ε, θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε αναλάβει και καλύτερες, πιο δραστικές λύσεις οι οποίε δεν θα βασίζονται στι εθνικέ κυβερνήσει, αλλά σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτή είναι μια ιδέα που θα μπορούσαμε να την εξετάσουμε. Εμεί ε, επικεντρωθήκαμε κυρίω στα, στα προγράμματα εγγύσεων των καταθέσεων και πώς αυτά τα προγράμματα μπορούν να ενισχυθούν και σε ό,τι αφορά τη συμβολή για την αντιμετώπιση των κρίσεων από τους ομίλους. Και επίσης σκεφτόμεθα και έτσι σε στα πλαίσια της αλληλεγγύης να συνδέσουμε όλα αυτά τα, τα προγράμματα εγγύησεων. Αυτό θα μπορούσε ίσως να δώσει ένα βαθμό συμβολής και από τον ιδιωτικό τομέα για τους διασυνοριακούς τραπεζικούς ομίλους. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια που περιγράφεται θα πήγαιναν προς την ίδια κατεύθυνση. θα είχαν και αυτά έτσι, την πτυχή της ε, παρέμβασης ώστε να καλύπτεται το κόστος αυτό της αντιμετώπισης της, έστω της πρώτης αντιμετώπισης της κρίσης από τους ιδιωτικούς φορείς. Σε ό,τι αφορά τώρα την σκοπιμότητα της χρήσης των ε, ε, ευρωπαϊκών κονδυλίων και πώς μπορούν ε, οι επιπλέον πόροι να χρησιμοποιηθούν από τα διάφορα κρατημέλη, ε, ως προς αυτό δεν μπορώ να σας δώσω ιδιαίτερη απάντηση. Αυτό όντω θα αποτελέσει πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Τώρα, για το κατά πόσο μπορούμε να έχουμε μια κεντρική υποπτική αρχή που θα δράσει συνδυασμό με τις εθνικές αρχές, αλλά όπου οι ε, εθνικές αρχές ε, θα έχουν εκχωρήσει εξουσία στην Ευρωπαϊκή Αρχή. Αυτό θα μπορούσε ίσως να αποτελέσει περαιτέρω διεύρυνση αυτού που τώρα συμβαίνει. Γιατί η νέα δομή των πραγμάτων ε, έχει και αυτή την πτυχή ε, ενσωματωμένη. Θα υπάρχει δηλαδή ένας κεντρικός φορέας που θα κάνει την ε, γενική εποπτεία και η καθημερινή εποπτεία θα γίνεται από τους ε, επόπτες των τραπεζών. Αλλά ένα κομμάτι των, ε, της υποπτίας θα γίνεται δυνάμει των κοινών κανόνων και της μεθοδολογίας που θα καθορίζει αυτή η κεντρική αρχή. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που γίνεται είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως μπορούμε να εξελίξουμε περισσότερο στο μέλλον. Thank you θέλεις το λόγο? Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Καρόζιο, εμείς δεν μιλούμε κάθε, μέρα σε αυτή την Επιτροπή για πρωτοβουλίες που προέρχονται από τις ε, πρωτεύουσε, αλλά αν δούμε πόση ανησυχία έχει δημιουργηθεί στις μεγάλες πρωτεύουσες αυτού του κόσμου όταν μιλούμε για τη ρύθμιση των τραπεζών, είτε είναι το Λονδίνο αυτό, είτε είναι η Ουάσιγκτον, είτε άλλες μεγάλες πρωτεύουσες, Παρίσι, τότε πραγματικά αναρωτιόμαστε αν εμείς με τις δικές μας ευρωπαϊκές προτάσεις παρουσιαζόμαστε να το παίζουμε λίγο έξυπνοι. Και η ανησυχία αυτή των μεγάλων πρωτευουσών του, του κόσμου δεν σχετίζεται άμεσα με τα προβλήματα αυτά που καταδεικνύουμε εμείς ότι δηλαδή δεν υπάρχει συγκεκριμένη μορφή ρύθμισης του τραπεζικού συστήματος. Υπάρχουν ως προς αυτό αρκετές προτάσεις διαφορετικές από όλο τον κόσμο, είτε για να εξασφαλίσουμε την, την ε, αξιοπιστία, είτε για να εξασφαλίσουμε την, τη βιωσιμότητα σε μακροπρόθεσμα, είτε για να έχουμε ρευστότητα, ε, για την παροχή κεφαλαίων, μιλούμε για αναγκαιότητα ασφαλιστικών συστημάτων των τραπεζών, παγκόσμιο σύστημα ασφαλιστικών συστημάτων τραπεζών. Ο Ομπάμα τώρα έκανε και μία έτσι πολύ επανεστατική πρόταση. Είπε, αφήστε να διαχωρίσουμε το τραπεζικό σύστημα για να κάνει το, τη δουλειά που πρέπει, την καθημερινή δουλειά που αφορά τους καθημερινούς πελάτες του. Όλες αυτές οι προτάσεις, εντάξει, πρέπει να αξιολογηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε ήδη εμείς μια στρατηγική και τι θεωρείτε εσείς πιο σημαντικό, εσείς πώς, πώς, βλέπετε αυτή την πρόταση να διαχωριστούν δηλαδή οι, οι τράπεζες και να αντιμετωπιστούν με διαφορετικούς κανόνες. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσουμε έτσι να συμπυκνώσουμε λιγάκι τις ερωτήσεις για να μπορέσει να απαντήσει και ο κύριος Καρόζιο. Αναφέρατε πολλές εκθέσεις που συζητούνται, ειδικά και στην FSB και στην Επιτροπή της Βασιλείας. Το φάσμα αυτό των διαφόρων παρεμβάσεων που αναφέρατε, όντως συζητείτε τώρα, Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις ως προς αυτό, ειδικά σε ό,τι αφορά τις ε, επαναστατικές ακραίες προτάσεις, να διαχωριστούν δηλαδή ε, οι, οι τράπεζες επενδύσεων από τις ε, υπόλοιπες χρηματοπιστωτικές τράπεζες με χρηματοπιστωτικά καθήκοντα, ας πούμε. Το θέμα που τίθεται εδώ είναι ότι ακόμη δεν είναι σαφές πώς αυτό θα συμβάλλει στο να αυξηθεί η σταθερότητα του δημοσιονομικού συστήματος. Ε, κάποιος διαχωρισμός του τύπου που προτείνετε εσείς ήδη είχε γίνει. Στη ΣΥΠΑ, α πούμε, υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι ξεχωριστέ οι επενδυτικέ τράπεζε από τι καταθετικές. Ε, Όπω θα έχετε δει, οι αρχέ στο τέλο είχαν να αντιμετωπίσουν πρόβλημα γιατί έπρεπε να διασώσουν και τις επενδυτικές τράπεζες γιατί η αποτυχία τέτοιων ομίλων δημιούργησε τεράστια προβλήματα στις οικονομικές αγορές και στις παραδοσιακές τράπεζες γιατί και αυτές επλήγησαν. Οπότε δεν είναι απόλυτα σαφές το πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό και από όσο ξέρω εγώ στις συζητήσεις που λαμβάνουμε μέρος αυτή η θέση έτυχε μικρή πλειοψηφία. Εν μέρη, ε, εκ μέρους εν μέρη ε, ακούστηκαν, ε, ε, υπερψηφίστηκε ας πούμε, από τις Βρετανικές αρχές, αλλά η δική μου ερμηνεία είναι ότι αυτή είναι μια συζήτηση που γίνεται, αλλά οι τελικές λεπτομέρειες δεν είναι διαθέσιμες για το ποια είναι δηλαδή η πρόταση. Αυτό που γίνεται τώρα σε σχέση με τις διάφορες ε, αλλαγές που γίνονται για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει είναι απαραίτητο. Είναι ένα βήμα που πρέπει να κάνουμε, είναι το πρώτο βήμα. Αυτές οι αλλαγές στις κεφαλαϊκές απαιτήσει θα επηρεάσουν και τη σύνθεση των δραστηριοτήτων των διαφόρων τραπεζών. χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, ε, ε, δομημένα προϊόντα, ε, επενδυτικές τράπεζες, όλοι αυτοί οι τομείς θα επηρεαστούν. Το κόστος λοιπόν κάποιων δραστηριοτήτων που ίσως να είναι αρκετά επικίνδυνες θα είναι πιο υψηλό. Οπότε αν θέλετε να κινηθείτε προς την κατεύθυνση αυτή, εντάξει, αλλά χωρίς να υπάρχουν φυσικά εμπόδια. Καλό θα ήταν να υπάρχει ένα σύστημα, ας πούμε, προοδευτικής φορολόγησης, αν μπορώ να το πω έτσι. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες προτάσεις που αφορούν και το μέγεθος των τραπεζών. Υπάρχει μια πρόταση πολύ δραστική που περιορίζει το μέγεθος μιας τράπεζας. Μπορεί δηλαδή να υπάρχει μεγάλο συγκεντρωτισμό ε, σε μια αγορά, να υπάρχει θέμα ανταγωνισμού. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα όμω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά τι ε, απαιτήσει, αντί να έχουμε συγκεκριμένο όριο, το οποίο δεν θα μπορούν να ξεπεράσουν οι τράπεζε ό,τι αφορά το μέγεθό του, θα μπορούσαμε να έχουμε μια κλιμακωτή φορολόγηση. Mm. Αυξημένε δηλαδή απαιτήσει για τι μεγάλε τράπεζε σύμφωνα με μια φόρμουλα που θα βρούμε. Right, colleagues, we've got our usual uh, position that... Συνάδελφοι, εάν ε, όλοι υποβάλλετε ερωτήσεις μακρηγορώντας όπως ο προλαλής σας, τότε δεν θα μπορέσουμε καν ε, να ολοκληρώσουμε τον πρώτο γύρο. Θα πρέπει ναι, ναι, ναι. να περιοριστείτε στο ένα λεπτό. Υποβάλλετε μία μόνο ερώτηση έτσι ώστε ο μιλητής να έχει τη δυνατότητα να απαντήσει. Θα έχουμε γύρους τριών ομιλητών, έτσι ώστε αν υπάρχουν επικαλύψεις να υπάρχουν άπαξ. Vicky Ford. Αλίσσα Φερέ ε, και Ντανούτα Χούμπνερ, η Βίκη. Quick, but I've got quite a few questions. Θα είμαι πολύ σύντομη. Σε σχέση με αυτή την ε, σοβαρή εργασία, μπορείτε να μας πείτε πώς έχει κατάσταση του προσωπικού. Ποιος αποφασίζει επίσης για τις ε, προδιαγραφές. Είπατε ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να αλλάξει τις ε, προδιαγραφές και ο, τελευταίος, ε, ο τελικός διαιτητής είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μιλήσατε για ολιστικές λύσεις σε σχέση με τις ε, ε, ανάγκες κεφαλαϊκών παροχών ως προς τις αποκαλύψεις το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Το IS 39 μπορεί να ισχύσει ως προς τη λογοδοσία. Ως προς το θέμα της ασφάλειας υπάρχει ένα θέμα δεοντολογίας ε, ως προς τους ε, κινδύνους και αυτό σημαίνει εξασφάλιση ε, όχι μόνο των μικροκαταθετών αλλά και των μεγάλων καταθετών. Πώς καλύπτονται όλα αυτά. Η Ελίσσα. Θα ήθελα να υποβάλω αρκετές ερωτήσεις. Πόσο μακριά κινηθήκατε ε, ως προς την κατανόηση ενός σημείου εκκίνησης εξάντε πριν αποτύχουμε θα πρέπει να μας απασχολήσει και η εναρμόνιση. Πιστεύετε ότι έχετε σαφή κατανόηση της κατανομής του βάρους μεταξύ διαφόρων αρχών τη στιγμή που υπάρχουν διατραπεζικές δραστηριότητες. Τρίτον, στο DGS θα πρέπει να κάνουμε πολλά, αλλά θα πρέπει να έχετε περισσότερες αρμοδιότητες έτσι ώστε να μην καταβάλει ο φορολογούμενος το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μπορεί λοιπόν αυτό να είναι ένα σαφές παράδειγμα για, τη, τα δικαιώματα των μετόχων, δηλαδή πώς μπορούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα πριν να ανακύψουν πραγματικά στην αγορά. Τενότα Χούμπνερ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της διαμεθεωριακής διαχείρισης που έθεσαν και άλλοι δύο συνάδελφοι, αλλά που είναι σημαντικό γιατί η Κομισιόν δεν έθεσε πραγματικά αυτό το πρόβλημα, ούτε πρότεινε λύσεις. Ερωτώ λοιπόν, μέχρι πού πιστεύετε ότι πρέπει να πάμε για να καθορίσουμε δεσμευτικούς κανόνες σε περίπτωση πτωχεύσεων, γιατί αν δεν υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες και υποχρεωτικές λύσεις, τότε δεν ξέρω τι βάρος πρέπει να δώσουμε στην πολιτική πτυχή που σημαίνει ότι τα κράτη θα χορηγήσουν ρευστά στους πεπτωχευμένους οργανισμούς. Μέχρι πού λοιπόν μπορούμε να το πάμε. Τι μπορούν να κάνουν οι εποπτικές αρχές. Εμείς πού θα θέσουμε τον πύχη. Yes, um, try to come in at sort of about four minutes. Ναι, παρακαλώ να περιορίζεστε στο τετράλεπτο. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά να. Ε, μάλιστα, εμείς ε, προβλέπουμε αύξηση του προσωπικού από 20 που έχει τώρα η γραμματεία σε 90 σε 4 χρόνια. Είναι σημαντική ποσοστιαία αύξηση, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι τεράστιο προσωπικό. Τώρα, για τη διαδικασία έγκρισης σας επιβεβαιώνω ότι σωστά καταλάβατε αυτά που είχα πει για τις υπερβολικές αναλήψεις κινδύνου από τράπεζες. Νομίζω ότι και που είπατε ότι μπορεί να αυξηθεί αν ε, επιχορηγούνται ή αν υπάρξει κάποιο ταμείο. Εγώ θα έλεγα ότι η ηθική κίνδυνη ε, είναι κάτι που πια δεν αποφεύγεται γιατί οι κυβερνήσεις έχουν θελήσει και για πολύ σωστούς λόγους να βοηθήσουν ε, τεράστιους δημοσιονομικούς ομίλους και η αγορά αναμένει κάτι ανάλογο να γίνει και στο μέλλον σε περίπτωση προβλήματος. Άρα νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να ταχθεί κατά μιας λύσης μόνο και μόνο επειδή θα δημιουργηθεί κάποιος περισσότερος ηθικός λεγόμενος κίνδυνος, αλλά πρέπει να δούμε πώς η χρηματοδότηση θα μπορούσε να λειτουργήσει σε συγκεκριμένους όρους, δηλαδή πώς, με ποιους κανόνες θα μπορούσαν οι πόροι αυτοί να χρησιμοποιηθούν από τους τραπεζικούς ομίλους που θα τους χρειαστούν. Πράγμα που συνδέεται με το άλλο θέμα του σε ποιο σημείο θα αποφασίζουμε, σε ποια ακριβή χρονική στιγμή ότι μπορούμε να παρέμβουμε. Ούτε χρήσιμο είναι ούτε δυνατόν νομίζω να υπάρχουν τέτοιοι αυτόματοι μηχανισμοί. Γιατί ακόμη και τα παραδείγματα που δίνουμε συνήθως όπως της του Αμερικανικού νομοσχεδίου Prompt Directive Action δείχνει ότι ιδιαίτερα για τις πολύ μεγάλες τράπεζες δεν μπορεί να υπάρχει αυτόματος μηχανισμός παρέμβασης. Γι' αυτό θα έλεγα ότι ο μόνος δυνατός τρόπος να λυθεί το πρόβλημα είναι οι επόπτες του συγκεκριμένου ομίλου να αξιολογούν συνεχώς τις συνθήκες και εκείνοι να αποφασίζουν ποια στιγμή θα έπρεπε να υπάρξει παρέμβαση. Πράγμα το οποίο φυσικά συνδέεται και με το κατά πόσον είναι αποτελεσματικό το κολέγιο των εποπτών ενός ομίλου. Εμείς προσπαθούμε να αυξήσουμε τον αριθμό και των κολεγίων και να διασφαλίσουμε ότι ακριβώς η λειτουργία τους θα συνίσταται σε κοινή αξιολόγηση του κινδύνου μεταξύ όλων των εποπτών ενός κολεγίου. Η FDIC τώρα και κατά πόσον θα μπορούσε να βελτιώσει τα πράγματα. Το πρόβλημα που τίθεται εδώ είναι Ποιες θα είναι οι σχετικές δικαιοδοσίες με, μεταξύ FDIC και εποπτών. Στις Ηνωμένε Πολιτείες υπάρχουν κοινέ δικαιοδοσίες, επικαλύπτονται κάπως, αλλά αυτό δημιουργεί και προβλήματα με αυτές τις επικαλύψεις. Διευκολύνεται μεν το ότι ανήκουν όλοι μαζί σε, στον ίδιο κρατικό οργανισμό, αλλά διαφέρει πολύ από το ευρωπαϊκό σύστημα όπου χρειάζονται και εθνικές και υπερεθνικές και τομεακές αρχές. Αυτό θα δημιουργούσε πολλά προβλήματα στην Ευρώπη. Πόσο δεσμευτικοί μπορούν να είναι οι κανόνες επιμερισμού του βάρους ή των βαρών εδώ μπορεί να υπάρξουν βέβαια μερικά γενικά κριτήρια για το ποιος θα ήταν ένας λογικός τρόπος καταμερισμού του βάρους και το επεξεργαζόμαστε αυτό, αλλά η μόνη πρακτική λύση θα ήταν να υποθέσουμε ότι υπάρχει μία ξεχωριστή και συγκεκριμένη λύση για κάθε όμιλο. Δηλαδή για κάθε τραπεζικό όμιλο να γίνεται μια κατά κάποιον τρόπο κατανομή εργασίας μεταξύ των αρχών και ως προς το τι δράση θα αναλάμβαναν και ως προς το τι πώς μάλλον θα χρηματοδοτούσαν σε περίπτωση επίγουσας ανάγκης. Τίποτε άλλο. Όχι τα εξάντλησα όλα. Μάλιστα. Οι επόμενοι τρεις ομιλητές. Ο Σβέν πρώτος. Κοιτάξτε, μία μόνο ερώτηση έχω. Όταν βλέπει κανείς τα προβλήματα εποπτείας των τραπεζών στην Ευρώπη, εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα της ευθύνης των κλάδων. Στις προτάσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, θεωρείτε ότι λύθηκε αυτό το πρόβλημα. Και δεύτερον, τι θα έπρεπε να γίνει κατ' για να λυθεί, αν δεν έχει λυθεί, για τις δικαιοδοσίες των κλάδων Α. Έπειτα, είπατε ότι πρέπει να συνδεθούν τα συστήματα εγγυήσεων στην Ευρώπη. Μερικοί όμιλοι έχουν μεγάλη παράδοση προγραμμάτων εγγύησης και επιτυχών, αλλά θα έπρεπε αυτά να καταστούν υποχρεωτικά ή θα δημιουργούνταν έτσι προβλήματα ανταγωνισμού μεταξύ ειδών τραπεζικής δραστηριότητας που μπορεί να μην είναι όλες ε, κοινού συμφέροντος όσο καλά και να έχουν λειτουργήσει στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Αυτό που μας απασχολεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να δούμε την πρώτη διασυνοριακή συνεργασία εποπτείας, διότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κοινοί κίνδυνοι και πρέπει να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη στο χρηματοοικονομικό σύστημά μας. Άρα η ερώτηση έχει ως εξή. Εάν θέλουμε να έχουμε ε, ευρωστία και νομιμότητα του συστήματος, καθώς και ασφάλεια, τότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη δύο στοιχεία Καταρχήν να έχουμε έγκαιρη προειδοποίηση, early warning, με ε, early tools, με έγκαιρους μηχανισμούς. Πιστεύετε ότι τα 27 κράτη-μέλη έχουν διορθωτικά μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να συγκριθούν. Δεν θα έπρεπε να βρούμε τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα τη στιγμή που συμμεριζόμαστε κοινού κινδύνους. Ευχαριστώ. Επειδή υπάρχει εποπτική αρχή, σημαίνει ότι το αντικείμενο εποπτείας μπορεί να τύχει εποπτείας. Ορισμένα προϊόντα που έχουν πολιθεί από τους ε, χρηματοπιστωτικούς φορείς είναι πολύ περίπλοκα προϊόντα και δεν γίνονται κατανοητά ούτε από αυτούς που τα πωλούν. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν περιορισμοί στα πολλούμενα προϊόντα. Αυτό ε, δεν θα διευκόλυνε τη δική σας εργασία. Δηλαδή, ως προς την ε, περιπλοκότητα των προϊόντων και την αποδοτικότητα της αγοράς, αυτό δεν έχει, αυτή η αιτιώδη συνάφεια δεν έχει καταδειχθεί και γι' αυτό θα ήθελα να εμβαθύνετε κάπως επί του θέματος θα πρέπει κανείς να έχει πολύ καλά επιχειρήματα υπέρ αυτής, ε, υπέρ της, υπέρ της ε, τάσης. Πρόκειται για ε, επιτροπή η οποία ασχολείται με τραπεζικά θέματα και όχι θέματα ασφαλείας. Well, to be honest, I think, um, Νομίζω το θέμα των υποκαταστημάτων θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ας δούμε το θέμα της Ισλανδίας, για παράδειγμα. Τις τράπεζες, δηλαδή, την τράπεζα μητέρα και τις θηγατρικές τράπεζες. θα πρέπει να αρκεστούμε στο, στην, στο αρχικό μας σχέδιο και να δούμε τις κεντρικές τράπεζες και τις διάφορες θηγατρικές στα διάφορα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην υπάρχουν δηλαδή προσκόμματα για εισδοχή από μια χώρα προέλευσης. Αλλά οι καταθέτες θα πρέπει να προστατεύονται οπουδήποτε κι αν βρίσκονται και σε οποιαδήποτε τράπεζα κι αν είναι πελάτες. Κάτι το οποίο δεν ίσχυσε στην ε, παρούσα περίπτωση. Δεν έχω μία λύση. Αλλά θα πρέπει να μας απασχολήσει η επάρκεια προστασίας προς τους ε, καταθέτες και του όλου συστήματος ε, εγκυοδοσίας των καταθέσεων που θα πρέπει να διέπει τις τράπεζες. Ως προς την ε, διασύνδεση των εγκυοδοτικών ταμείων καταθέσεων, εδώ έχουμε να κάνουμε σε, με διάφορες κατηγορίες τραπεζών μέσα στην ίδια χώρα. Αυτό θέλουμε να το συνδέσουμε δηλαδή τα, τις εγκαιοδοσίες καταθέσεων σε, στην ίδια χώρα και μεταξύ κρατών μελών. Θα πρέπει κανείς να διαθέτει βαρύ πυροβολικό, δηλαδή επαρκείς πόρους που να καλύπτουν τα ενδεχόμενα ατυχήματα και το κάθε εθνικό σχέδιο εγκαιοδοσίας καταθέσεων είναι μικρό σε σχέση με το μέγεθος της ε, αποτυχίας ε, ορισμένων μεγάλων τραπεζών. Αν δείτε όμως τη συνολική εικόνα των, ε, της κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε αυτή η δυσαναλογία δεν είναι και τόσο δραματική. Ως προς τα διορθωτικά μέσα και κατά πόσο υπάρχουν, ε, είναι παρόμοια και συγκρίσιμα, όχι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Προσπαθήσαμε να χαρτογραφήσουμε τους ε, διαφόρους μηχανισμούς εκεί που διατίθενται και τα αποτελέσματα είναι αποκαρδιωτικά. Υπάρχει μεγάλη απόκληση σε ορισμένες χώρες Υπάρχουν συστήματα ειδική διαχείρισης για να αντιμετωπίσει κανείς την κατάσταση μιας ε, τραπεζικής αποτυχίας. Σε άλλες χώρες δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και οι δικαστικές αρχές θα μπορούσαν μόνο να επιληφθούν του θέματος. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη ευρύτητα νομικών συστημάτων. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα πιο συνεπές σύστημα και συνεκτικό. οι κυβερνήσεις έπρεπε να προβούν σε διάσωση ομίλων σε μια κατάσταση κρίσης και το ζήσαμε αυτό. Γιατί διαφορετικά μια μερική επίλυση δεν θα ήταν ε, επαρκή στα πλαίσια ενός ομίλου ή μιας κοινοπραξίας. Αυτό αποκλείεται διότι έμπρακτα θα ήταν αδύνατον. Δηλαδή να υπάρχει μια συντονισμένη διαδικασία επίλυσης σε διάφορες χώρες. Αυτή η διαδικασία λοιπόν δεν αδυνατο δηλαδη να ενεργοποιηθεί και μειώνει τις εναλλακτικές που έχουμε ενώπιόν μας για παρέμβαση, ορισμένα προϊόντα είναι περίπλοκα και θα πρέπει να απαγορευτούν. Δεν είμαι αρμόδιος, διότι ως τραπεζικοί επόπτες ασχολούμαστε με τους άμεσους ή έμεσους κινδύνους που αναλαμβάνουν οι τράπεζες. Δεν έχουμε προβεί σε εποπτεία προϊόντων άρα δεν υπάρχουν κανόνες εποπτείας προϊόντων. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα έπρεπε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει περαιτέρω. Γιατί είναι δύσκολο να θέσει κανείς όρια για το τι μπορεί να γίνει στον τομέα της καινοτομίας και πολλές φορές είναι αδύνατο να αποφύγουμε την καινοτομία για να παρακάμψουμε τα όρια που θέτουμε. Από την άλλη πλευρά, πλευρά όμως, ίσως θα ήταν χρήσιμο να έχουμε μία τυποποίηση προϊόντων. Μία τυποποίηση λοιπόν η οποία θα πρέπει να τύχει ενθάρρυνσης η οποία μπορεί να έχει και δραστικό χαρακτήρα. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι ορισμένοι επενδυτές ίσως ε, περιοριστούν στη, στα προγράμματα επένδυσης. Άρα η τυποποίηση των προϊόντων θα πρέπει να προβούμε σε μία τυποποίηση των προϊόντων που, είναι, που μπορούν να ε, επιλεγούν για ορισμένες επενδύσεις τελικός γύρος. Όλα Σμιτ. Κύριε Κορόζιο, ίσως ε, θα πρέπει να απαγορεύσουμε τις μεγάλες τράπεζες. Με συγχωρείτε, λέει η πρόεδρος. Τα πηγαδάκια να απομακρυνθούν από την αίθουσα. Και αυτό περιλαμβάνει και τους ίδιους τους ε, βουλευτές και πρωτίστως αυτούς θα πρέπει να ξαναρχίσεις όλα. Κύριε Κορόζιο, στη χώρα μου αντιμετωπίζουμε ή αντιμετωπίσαμε ένα πρόβλημα ε, με τράπεζες που ήταν πολύ μικρές για να επιβιώσουν. Τώρα είναι πολύ μεγάλες για να αποτύχουν. Ναι. Αυτό θα πρέπει να είναι το ερώτημα. Ίσως θα πρέπει να απαγορεύσουμε την δραστηριότητα μεγάλων τραπεζών. Και αυτό συνδέεται με αυτό που κάνετε. Έχουμε 44 τράπεζες που δρούν διασυνοριακά, γύρω στις 40 αν δεν κάνω λάθος. Ε, ευεργέτησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δράση του στάθηκε ευεργετική. Καλημέρα σας. Όσοι εισηγήτρια του κιμέν για τους συστημικούς κινδύνους θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής θα ε, λάβετε υπόψη την έκθεση Rosière η οποία σημαίνει θα πρέπει μετά από τους κινδύνους και τον εντοπισμό τους να προβούμε και σε δράση. Εσείς θα βρισκόσαστε στη, σε όλα αυτά υποπτικά όργανα. Τι θα γίνει με τις κατευθυντήριες γραμμές που δεν είναι δεσμευτικές. Edward. σε εθνικό επίπεδο αρκούμαστε στην αποτελεσματικότητα των ε, τραπεζικών εποπτών. Πολλές φορές υπάρχουν ε, ειδικά θεσμικά όργανα από αυτού. Έχουν γίνει μελέτες για να συγκρίνουμε τις δύο τάσεις, διότι μέχρι τώρα ήμασταν ε, ουδέτεροι επί του θέματος. So Edward, can you, can you just sort of reiterate that? Μπορείς να επαναλάβεις. Um, Όχι, μιλάω για διαφορετικά μοντέλα που υπάρχουν στις διάφορες χώρες για την εποπτεία των τραπεζών. Στο, το FSA κάνει την εποπτεία στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάποια, σε κάποιες χώρες την κάνει η Κεντρική Τράπεζα. Μέχρι τώρα δεν έχουμε ακούσει κάτι, εκτός από κάποια δημοσιεύματα σε εφημερίδες. Υπάρχει κάποια έγκριση, κάποια ε, σύγκριση, συγγνώμη, κάποια έρευνα επίσημη, ότι ας πούμε η εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας έχει υπάρξει καλύτερη, πιο αποτελεσματική από την εποπτεία από άλλους φορείς. Quickly, um, has there been any benefit? Αν έχει υπάρξει όφελος από τις διασυνοριακές δραστηριότητες των τραπεζών. Ναι, θα έλεγα εγώ. Εντάξει, εγώ μπορώ να μιλώ βέβαια εκ, εξ ονόματος και των εθνικών ε, ποπτών, αλλά έχει αυξηθεί ο ανταγωνισμός που προέρχεται από χώρες, από άλλες χώρες. Και η ποιότητα επίσης των τραπεζών που δρούν διασυνοριακά έχει επίσης βελτιωθεί. Και γενικότερα ε, δεν μπορούμε να έχουμε ολοκληρωμένες αγορές χωρίς επιχειρήσεις που να περνούν τα σύνορα και να, παράσχουν, και να παρέχουν α, υπηρεσίες. Τώρα, οι κατευθυντήρες γραμμές και αν θα είναι δεσμευτικές ή όχι. Νομίζω ότι είναι περίπλοκο το θέμα αυτό. Δηλαδή, ποια είναι η σχέση μεταξύ του, της ΕΤΕ και των νέων ε, εποπτικών αρχών. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αναλύσουμε βαθύτερα μάλλον δεν θα ήταν χρήσιμο να προσθέσουμε και άλλα νομοθετικά κείμενα και άλλες νομοθετικές απαιτήσεις, γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό είναι θέμα του πώς θα γίνει πρακτικά η ολοκλήρωση. Και αυτό θα το δούμε. Υπάρχουν παραδείγματα συνεργασίας που ήδη γίνεται σε ένα βαθμό, ας πούμε τα stress test που σας ανέφερα πιο πριν κάτι δηλαδή που γίνεται χρησιμοποιώντας τις αναλύσεις και τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα διάφορα σενάρια που πρέπει να μελετηθούν. Και αυτό μετά περνάει στους επόπτες που εφαρμόζουν τα σενάρια αυτά στις ε, ε, τράπεζες και κάνουν την αξιολόγηση επιπτώσεων και μετά με βάση αυτή, την, αυτή η αξιολόγηση μάλλον επιπτώσεων μπαίνει, γυρίζει πίσω στην μακροαξιολόγηση των συνεπειών. Συζητούμε λοιπόν και στρατηγικές εξόδου, όπου υπάρχει και πάλι σύνδεσμος των ε, μακρομέτρων και των συνθήκων που υπάρχουν στις διάφορες ε, τράπεζες, δηλαδή αν είναι αρκετά δυνατές για να υποστηρίξουν και να συνεχίσουν να υπάρχουν ή αν θα πρέπει να αποσυρθούν. Είναι περίπλοκο το σύστημα. Και νομίζω ότι πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό καλύτερα. Τώρα, για το ποιο μοντέλο είναι καλύτερο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ε, επίσημες έρευνες, μελέτες. Ε, έχουν γίνει πολλές ακαδημαϊκές έρευνες και από όσο ξέρω είναι δύσκολο να αποδείξει κανείς έτσι με στατιστικό ας πούμε τρόπο ε, ποιο μοντέλο είναι καλύτερο και πιο αποτελεσματικό. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι Υπάρχει μια τάση στην Ευρώπη, τελευταίος, προς ένα μοντέλο δι, διτό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ας πούμε στην, στη Γαλλία και στην Ισπανία, στην Ολλανδία ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, αυτή η τάση. Okay, thank you very much. Um, we've, we've come to... Ωραία έληξαν όλοι οι γύροι. Θα είχαμε σωρία ερωτήσεων βεβαίως. Ποτέ δεν μας αρκεί ο χρόνος. Σας ευχαριστούμε θερμά και είστε πάντα ευπρόσδεκτος εδώ, στο εγγύς μέλλον και όχι στο μακρινό ή δυνατόν. Συνάδελφοι, προχωρούμε. We need move on to the exchange of απόψεων τώρα. Δεν έχουμε χρόνο για ιδιωτικές συζητησούλες, γιατί αρχίσαμε αργότερα. Γιατί δεν είχαμε απαρτία. Τώρα θα προβούμε στη δεύτερη ανταλλαγή απόψεων, στο CRT3. Μίλησα με τον εισηγητή και ίσως θα ήταν σκόπιμο η Κομισιόν να μας απαντήσει μέχρι το τέλος της συζήτησης. Δίνω το λόγο στην Αρλίν για να παρουσιάσει αυτή τη συζήτηση. Σας παρακαλώ σταματήστε τις συζητησούλες. We'll do it to you when it's your report, so stop. Θα το κάνουμε σε σας όταν παρουσιάζετε δική σας έκθεση, Αρλίν. Um, Χαίρομαι διότι μου δίνετε τη δυνατότητα αυτής της συζήτησης, ε, διότι δεν προηγήθηκε, ούτε είχαμε και την Κομισιόν μαζί μας. Άρα αρχίζουμε εκ του μηδενός. Αλλά βεβαίως η χρηματοπιστωτική κρίση οδήγησε σε μια γενικότερη συζήτηση ως προς τις τράπεζες, τους ε, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και βεβαίως και τα μπόνους των ε, στελεχών των τραπεζών. Γι' αυτό έχουμε αυτή την πρόταση CRD3. Θα θέλαμε να αντιμετωπίσουμε μελλοντικές ενδεχόμενες κρίσεις στον τραπεζικό τομέα, να μην αναλαμβάνονται κίνδυνοι που οδηγούν σε ε, σε μεγάλες απώλειες και νομίζω ότι οι φορολογούμενοι δεν είναι υπεύθυνοι για την ε, επιβίωση των τραπέζων. Μιλάμε για 5,33 εκατομμύρια επιδότηση διευρωπαϊκά για τις τράπεζες, δηλαδή το αντίστοιχο του ΑΕΠ της Γερμανίας. Μιλάμε για πολύ μεγάλα αριθμητικά στοιχεία που θα πρέπει να μην μας απασχολήσουν στο μέλλον. Επίσης, θα πρέπει να δούμε και τα μπόνους των στελεχών των τραπεζών. Τα συστήματα ή τα διαρθρωτικά μέτρα θα πρέπει να τίθενται σε ορθολογική βάση έτσι ώστε να ε, να υπάρχει ένα αντίτιμο στην απόδοση αλλά να μην είναι υπέρμετρη αυτή η απόδοση, η άδικη. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς ως προς ε, ένα τύπο νομοθετήματος που διέπει τον τραπεζικό τομέα. Ακούσαμε την πρόταση ε, Ομπάμα σε σχέση με τα hedge funds να περιορίσουμε το μέγεθος των τραπεζών. Είχαμε σοβαρές συζητήσεις ως προς ένα ειδικό τέλος ή φόρο, διατραπεζικό φόρο μιλάμε για ασφαλιστικά σχέδια, όλα αυτά συζητώνται. Επίσης, στις ακροάσεις της είπαμε, είδαμε πώς εξελίχθηκε το ζήτημα ως προς την ε, διατραπεζική κρίση και στον Ταβό στο τέλος της εβδομάδας η μεταρρύθμιση των τραπεζών και το θέμα των ε, αμοιβών θα τεθεί επιτάπητος διότι θα χρειαστεί διαρθρωτική μεταρρύθμιση στον εθνικό τομέα από τότε που προωθήθηκε αυτή, τη, αυτή η τάση υπάρχουν υπερισφορές στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία. Επίσης ε, μιλάμε για αποζημιώσεις της τάξης του, 1, του 1 εκατομμυρίου pounds. Το ίδιο προώθησε και η τράπεζα Barclays Δηλαδή υπάρχουν και μεταφερόμενα μπόνους 100% για μία τριετή περίοδο. Αυτά τα αναφέρω διότι το υπόβαθρο αυτής της οδηγίας μας δείχνει ότι υπάρχει μία εξελικτική πορεία ως προς ε, ε, ορισμένα ερωτήματα που θα ήθελα να επαναφέρω. Θα ήθελα η Κομισιόν και τα μέλη να απαντήσουν δεν διατρέχουμε κινδύνους με αυτή την οδηγία. Και οι άλλες ad hoc οδηγίες απαντούν στους κανόνες της Βασιλείας ως προς τη τραπεζική εποπτεία. Τέλος, μιλάμε για ένα νομοθέτημα το οποίο ε, αντί να μας ωφελεί μακροχρόνια είναι απαρχαιωμένο πλαίσιο. Θα θέλατε λοιπόν να προωθήσουμε ad hoc λύσεις παρά να έχουμε μία άρδιν μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα. Μου φαίνεται ότι η προσέγγιση μας είναι μία προσέγγιση ad hoc σε σχέση με το τι συμβαίνει στη Βασίλη. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουμε ηγετικό ρόλο στη, στα διεθνή φόρα παρά να έχουμε στάση αναμονή στη Βασιλεία για να δούμε τι θα συμβεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε ουραγοί μια ζωή. Πολλές φορές είχαμε ηγετικό ρόλο σε άλλα θέματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι και ριζοσπαστικοί. Έχουμε, απο, έχουμε απόψεις και ιδέες δεν ανταποκρινόμαστε μόνο στα παγκόσμια τεκτενόμενα. Με αυτή την νομοθεσία θα πρέπει να διασφαλίσουμε κανόνες που να μας υπηρετούν μακροχρόνια, όχι μόνο για τα επόμενα έτη και να επανέλθουμε, να ξαναμεταρρυθμίσουμε το όλο Θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν πώς ε, ανταποκρινόμαστε στις αλλαγές της ε, Βασιλείας. Σε αυτή την πρόταση έχουμε να κάνουμε με τρεις συνιστώσεις ε, κεφαλαιακές ε, απαιτήσει για το διατραπεζικό τομέα, το θέμα των αμοιβών και το οποίο είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Θα πρέπει να δούμε τι κάνανε οι τράπεζες στο παρελθόν. Στο ε, παρελθόν δεν υπήρχαν εθνικά σχέδια διάσωσης από τις κυβερνήσεις. Δεν περίμεναν κάτι τέτοιο οι τράπεζες. Τον 19ο αιώνα στις ΗΠΑ ή στη Βρετανία ε, έπρεπε να προωθούσαν ένα equity buffer το οποίο να ήταν 25% της ε, συνολικής ρευστότητας. Και όσο υπάρχει μεγαλύτερη προστασία, υπάρχει μείωση αυτών των προαπαιτήσεων. Και τέλος, οι τράπεζες είχαν ένα 3% των περιουσιακών στοιχείων ρευστοποιημένο ή μία ολική ρευστοποίηση της τάξης του 10%. Δεν λέω ότι θα πρέπει να κινηθούμε, να παλινοδίσουμε στο 19ο αιώνα, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους. Ο Άντρου Χάλντεϊν της Τράπεζας της Αγγλίας πρότεινε να ξαναβρεθούμε στο 1360 όπου ένας κεντρικός τραπεζίτης εκτελέστηκε δημοσία επειδή δεν ανταποκρίθηκε στο καθήκον του. Το κοινό δεν θεωρεί ότι θα πρέπει το κέρδος να ιδιωτικοποιείται, αλλά θα πρέπει να υπάρχει κοινωνικοποίηση των ζημιών. Το θέμα των αμοιβών θα πρέπει να μας απασχολεί, θα πρέπει να δούμε τι αντισταθμίσεις υπάρχουν. Θέλουμε ένα σταθερό τραπεζικό σύστημα, να υπάρχει επαρκές κεφάλαιο πίσω από τις τράπεζες, να, να, διοδοτούν, να δανειοδοτούν οι τράπεζες. Άρα θα πρέπει να δούμε τι αντισταθμίσματα υπάρχουν στο τομέα της ασφαλείας. Θα πρέπει να υπάρχει ε, καλύτερη κεφαλαιοποίηση δηλαδή των τραπεζών. Η Βασιλεία ορίζει ορισμένους κανόνες. Μιλάμε για μια πολιτική ε, ως προς μετοχές, για τιτλοποίηση και χρειάζεται correlation trading. Τώρα υπάρχει ένα κατόφλι για το correlation trading, αλλά βασιζόμαστε στη βασιλεία. και είχαμε και ένα έγγραφο διαβούλευσης από τη Βασίλεια για τα όρια ε, το, του, του σορευτικού αυτού καθεστώτος, κατά πόσο το αρχικό κεφάλαιο είναι υγιές κεφάλαιο και ποια είναι τα σορευτικά ε, στρεβλωτικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Δεν έχουμε τελικές θέσεις, αλλά πώς θεωρεί η Κομισιόν ότι μπορούμε να ενσωματώσουμε αυτές τις αλλαγές στη οδηγία και ε, αν ε, αλλάξει το ποσοστό, ε, το ποστό μόχλευσης, πώς θεωρείτε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το όλο ζήτημα γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν ε, φτωχεύσουν οι Lehman Brothers είχαν μία αναλογία ενός 11% κεφαλαίου σε σχέση με το συνολικό κεφάλαιο που θα έπρεπε να διέθετα. Κατά το τέλος του 2010 ή ε, Ιανουάριο 2011 θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο έτσι λέει η Κομισιόν και το Συμβούλιο, έχει μεγάλη σημασία ο ρυθμός δανειοδότησης και βεβαίως ένα φορολογικό καθεστώς. Και εάν οι τράπεζες έχουν χρήματα για πόνους, τότε δεν λείπει το κεφάλαιο. πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με το grandfathering των περιουσιακών στοιχείων και στο θέμα της τιτλοποίησης θεωρούμε ότι η τιτλοποίηση, η επανατιτλοποίηση δεν είναι ο πυρήνας, δεν αποτελούν τον πυρήνα της κρίσης. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τα χρεόγραφα πώς θα ορίσουμε την επανατιτλοποίηση, αλλά υπάρχουν και θέματα που δεν έχουμε ορίσει σε σχέση με περίπλοκες επανατιτλοποίησεις. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι πολυσχηδείς επανατιτλοποιήσεις θα πρέπει να εποπτεύονται από ε, συγκεκριμένες εποπτικές αρχές και ποιες θα είναι οι εισφορές στα τέλη που θα ισχύουν σε αυτή την περίπτωση. Το Συμβούλιο δεν το δέχτηκε αυτό γιατί θεώρησε ότι είναι ε, ένα επαχθές πλαίσιο για τις εποπτικές αρχές, διότι είναι πολύ υψηλό το κόστος των τίτλοποιήσεων ή των επανατίτλοποιήσεων. Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε δεν υπάρχει υψηλός βαθμός ε, επικινδυνότητας. και δεν θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχο κεφάλαιο κάλυψης αυτών των κινδύνων. Τι εννοεί η Επιτροπή όταν μιλάει για ε, πολυσχήδη επανατιτλοποίηση. Τώρα, ως προς αμοιβέ, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα κινηθούμε με βάση την αρχή business as usual. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία διότι οι τράπεζες είχαν μεγάλα κέρδη από τις κρατικές επιδοτήσεις, γιατί υπήρχαν χαμηλά επιτόκια, δεν υπήρχε ανταγωνισμός 150 δισεκατομμύρια ήταν τα κέρδη της Wall Street. Το ίδιο ισχύει και για το City του Λονδίνου. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε τους κανόνες που μας διέπουν, χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια και να μην υπάρχει αυτός ο, ο δεσμός μεταξύ αμοιβών και μπόνους και ανάληψης κινδύνου. Το Συμβούλιο ε, έλαβε υπόψη το Pittsburgh και το, τους G20 για να υπάρχουν ελάχιστες ε, προδιαγραφές για μεταβλητές αμοιβέ ανάλογα με το προφίλ των τραπεζών. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ε, μακροχρόνια αποδοτικότητα, να μην υπάρχουν εγγυημένα πόνους, και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το εξής. Γιατί γιατί υπάρχουν σχέδια, κρατικά σχέδια διάσωσης τα οποία προωθούνται και παρόλα αυτά οι τράπεζες δεν κόβουν τα ε, μπόνους και τις υπέρογγες αμοιβέ. Το 50% κάθε μπόνους θα πρέπει να χορηγείται σε χρεόγραφα και όχι σε ρευστό να μην υπάρχει υψηλή ανάληψη κινδύνου, μεγάλη ε, ανάληψη κινδύνου, να υπάρχει ένα spread του bonus σε μία τριετία. Και δεν ξέρω τι εννοούμε όταν λέμε υψηλά bonus. Και θα πρέπει να υπάρχει μεταφορά bonus ανάλογα με την αποδοτικότητα. Δηλαδή όταν χαμηλώνει να χαμηλώνουν και τα bonus. Ορισμένες ε, κυβερνήσεις ε, προχώρησαν περισσότερο από το FSB. Στο Ηνωμένο Βασίλειο το δύο, τα δύο τρίτα των πόνους ε, μεταφέρονται σε μία τριετία. Αυτό αφορά και την Αγγλία και την Ολλανδία. Δηλαδή έχουμε πακέτα αμοιβών και δεν μπορούμε να δεχτούμε τα πόνους να είναι υψηλότερα από τις αμοιβέ και εν περιπτώσει δεν υπάρχουν ε, ρητές υποχρώσεις. Επίσης θα πρέπει σε ένα bonus pool να υπάρχει μια συγκεκριμένη φορολόγηση. Γίνονται ακροάσεις και στις ΕΠΑ που ίσως ενταχθούν στην ε, πρόταση FSP. Θα δούμε τι θα γίνει το Μάρτιο την Άνοιξη γενικότερα, θέλουμε να αναλάβουμε αυτό τον κίνδυνο, δηλαδή να ε, λάβουμε νομοθετικά μέτρα τα οποία να είναι στο τέλος απαρχαιωμένα, πριν καν θεσμοθετηθούν. Η τριετής περίοδος αναπομπής είναι ε, σωστή γιατί υπάρχουν πιστοτικοί κύκλοι που είναι πολύ μεγαλύτεροι το 50% των αμοιβών είναι ε, λογικό. έτσι ώστε να υπάρχει σωστή απορρόφηση κεφαλαίου. Γιατί οι αμοιβέ δεν πρέπει να καταβάλλονται ε, μόνο με βάση τα μερίσματα, ούτε θα πρέπει να είναι 100% σε μετοχές τι θα γίνει με τις τράπεζες που έλαβαν κρατική βοήθεια. Θα πρέπει να διασώζουμε τράπεζες. Αν διασώζονται θα πρέπει να έχουν ειδικού κανόνες. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα πρέπει να επανειδωθεί το θέμα του, των πόνους. Επίσης θα πρέπει να ενδυναμώσουμε την διαφάνεια σε σχέση με την καταβολή μπόνους. Δηλαδή υπάρχει σύνδεσμος μεταξύ επικίνδυνων δραστηριοτήτων, δραστηριοτήτων κινδύνου και αμυφής. Τι μπόνους ε, λαμβάνουν τα στελέχη, θα πρέπει να υπάρχουν στους ετήσιους ε, ισολογισμούς και επίσης οι μέτοχοι θα πρέπει να έχουν μια σαφή ιδέα για την πολιτική αμοιβών. Ως προς τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβιάσεων, πώς θα πρέπει να καλύπτεται το όλο ζήτημα. Έθεσα σωρία ερωτημάτων, δεν έδωσα καμία απάντηση, αλλά με τη συζήτηση θα γίνει αυτό. Και αυτό θέλω να γίνει πριν αρχίσω την συγγραφική μου δραστηριότητα, γιατί αυτή δεν ήταν παρά η προφορική. Α, σας ευχαριστώ. Κάποτε θα έχουμε το χρόνο, ελπίζω, να τα συζητήσουμε και πιο λεπτομεριακά. Είμαστε και αύριο εδώ βέβαια. Λοιπόν, θα ήθελα να κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών. Jean-Paul Gauzes, Peter Skinner, Wolf Klintz and myself. And I then want to go... I, I, yes, okay. So we now want... You do have to signal even if you're a shadow. Uh, Pascal Canvin, anybody else? Right. Um, I might try to... Κανείς άλλος, καμία άλλη. προς το παρόν τα πάμε όλα καλά σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Βίκη. Είμαι και σκιώδης, άρα θα μπορείς να με βγάλεις από τον κατάλογο των σκιωδών. Α, ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια. Και εγώ ήθελα, ευχαριστήθηκα που είδα ότι πολλά από αυτά που είχα ζητήσει την προηγούμενη φορά τα έλαβε υπόψη. Ιδιαίτερα το ότι δεν πρέπει συστηματικά οι φορολογούμενοι και οι φορολογούμενες να πληρώνουν την ύφη που αποτελούν οι τράπεζες. Επίσης, έλαβε υπόψη και άλλες συζητήσεις που γίνανε τις περασμένες δέκα μέρες και με τους Αμερικανούς και τις Αμερικανίδες. Γιατί εδώ το θέμα είναι σφαιρικό το πρόβλημα. Λοιπόν, Ο φόρος συνυπευθυνότητας που, για τον οποίο μίλησε ο Ομπάμα ίσως θα ήταν χρήσιμη ιδέα να συζητηθεί και από εμά, αλλά βέβαια να το δει η Επιτροπή αυτό η Κομισιόν. για να φανεί έτσι ότι δεν ε, μένουμε πίσω στις νομοθετικές μας προτάσεις. Λοιπόν, συμφωνώ ότι Από την τελευταία φορά που τα είπαμε, η διατύπωση του εγγράφου ίσως δεν έλεγε αρκετά για τα μέτρα που θα έπρεπε ή θα ήθελαν να λάβουν οι κυβερνήσεις και το πρωί ήδη συζήτησα με ορισμένους τα τραπεζικά και κατάλαβα ότι ορισμένες χώρες μέλη προτίθενται να λάβουν μέτρα υψηλότερου επίπεδου από αυτά που προτείνονται επισήμως και πανενωσιακώς. Πράγματι μπορεί μερικές χώρες να θέλουν να ανεβάσουν τον πύχη ψηλότερα. Προς στιγμήν η διατύπωση θα μπορούσε να καταστήσει δύσκολο για, ορισμένα, για οποιοδήποτε κράτος να ξεπεράσει τον ενωσιακό πύχη και πρέπει αυτό να το διορθώσουμε για το λεγόμενο correlation trading έχω μπερδέψει τα αρχικά τώρα το QIS είναι το, η αξιολόγηση της βασιλείας κάτι τέτοιο το έγγραφο είναι πάνω από 150 σελίδες και γι' αυτό δεν πρόλαβα να το τελειώσω η τελική του μορφή θα εκδοθεί τον Ιούνιο τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία για αυτά τα θέματα που ακόμη τα επεξεργάζονται. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε εγκρίνουμε ένα τμήμα και θα επανέλθουμε, δεν ξέρω ποια είναι ακριβώς η σωστότερη μορφή. Αλλά ακούσαμε και πριν από τον πρόεδρο της ΕΑΕΤΕ ότι οι Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες πρέπει μέχρι το 2011, δηλαδή στην ουσία μέχρι τα τέλη του φετινού χρόνου για να ετοιμαστεί κάτι το 12 να έχουν ήδη εγκρίνει προτάσεις για αυτό θα το δούμε Σε ευχαριστώ επίσης για το θέμα του grandfathering της παππουδοποιήσεως. Αφού μιλάμε για κεφάλαια μέχρι το 4% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ, είναι πολύ εκφοβιστικός αριθμός αυτός. Αλλά τέλος πάντων θα τα δούμε στην αξιολόγηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες αντιμετωπίζονται μέσα στο κείμενό σου. Είναι σωστό λοιπόν να έχουμε κάποιους ε, κανόνες στους οποίους να πρέπει να, ε, τους οποίους πρέπει να τηρούν. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ και, για τις, και στις εκθέσεις, γιατί έχω την εντύπωση ότι στην τρίτη σελίδα υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα, περισσότερα από έχουν ξεκαθαριστεί. Υπάρχουν τρεις αιτίε για αυτά τα εκρέμη ερωτήματα. Καταρχήν το χρονοδιάγραμμα. Εφαρμόζουμε την Βασιλεία 2, συζητούμε το CAD3, προετοιμάζουμε το CAD4, συζητάμε για το CAD5 και πίσω από την κοινοβουλευτική συζήτηση μιλούμε και για, την, ε, ε, για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την Επιτροπή της ε, Βασιλείας. Είμαστε στο CAD3. Έχουμε την, τη Βασιλεία και, για το ίδιο κεφάλαιο και το CID 4 και μας μένει εκρεμές το CID 5 Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα δούμε από κοινού. Τελικά τι ακριβώς θέλουμε και τι πρέπει να γίνει και μέχρι πότε και πώς θα καταφέρουμε να έχουμε μια χρονικώς σωστή διαχείριση, τουλάχιστον ε, σε πολιτικό επίπεδο, σε ό,τι αφορά την, την ε, Επιτροπή της Βασιλείας. Για να μην ε, αντιδρούμε πάντα κατόπιν εορτής. Και επίσης, χρονική σύμπτωση με την με τη Βασιλεία. Αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό. Και επίσης έχω την άποψη, όπως και πολλοί άλλοι, ότι η εφαρμογή του CD3, όπως έχει τώρα, μέχρι το τέλος του έτους, μάλλον είναι πολύ νωρίς για να ολοκληρωθεί. Εμείς μέχρι τότε θα μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτό για το οποίο θα έχουμε τα συγκεκριμένα δεδομένα. Και εκεί ε, είναι που δεν έχουμε συγκεκριμένες μελέτες και μάλλον πρέπει να συνδέσουμε το CD3 με το CD4. Χρειαζόμαστε δηλαδή μια συνολική εποπτεία εικόνα των πραγμάτων. Ε, τώρα η προσαρμογή ε, για, ε, την επανατιτλοποίηση πρέπει να διευρυνθεί. Στην τελευταία ε, οδηγία για τις τράπεζες είχαμε ζητήσει από την Κομισιόν να εξετάσει τι γίνεται με την εφαρμογή του G20 και της Βασιλείας, τι σημαίνουν όλα αυτά και αν, τι γίνεται με την, υψηλότερη θέση, με την, θέση, με την θέσπιση υψηλότερων α, συντελεστών. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει απάντηση από την Κομισιόν. Η αξιολόγηση λοιπόν του κινδύνου είναι απαραίτητη. το θέμα πρέπει να, ε, συνεχίσει, να, συνεχίσουμε να το μελετούμε. Επανατιτλοποιήσεις, μπορούν να θεωρήσουμε ότι είναι μια, ένα πρόβλημα, που, μια αιτία της ε, κρίσης και πρέπει να δούμε όλα αυτά και στα πλαίσια της διαφάνειας. Επίσης πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι γίνεται με αυτή την ε, ε, ιδιαίτερα περίπλοκη τιτλοποίηση. Να ξέρουμε δηλαδή τι ακριβώς σημαίνει αυτός ο όρος. Μήπως θα πρέπει να τον διαγράψουμε τελείως και αν δεν γίνεται έλεγχο εποπτικός, εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ. Πρέπει να υπάρχει σαφή και αυστηρός έλεγχο. Τα μπόνους τώρα δεν μπορούμε να τα δούμε ανεξαρτητά από τις αποδόσεις. Το βασικό σημείο όμως είναι η βάση ε, ε, μέτρησης. Ποια είναι η βάση για τα μπόνους που δίδονται. Και αν υπάρχει μπόνους θα πρέπει να υπάρχει και μάλους σε περίπτωση αντίθετη. Να υπάρχει δηλαδή αντιστοιχεία. Και αυτό θα πρέπει να γίνει πάλι με βάση την ε, βάση επιλογισμού, η οποία θα πρέπει να είναι διαφανής. Επίσης, θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με την ευρωπαϊκή δομή των ε, ε, τραπεζών. Το να φορτώνουμε τις τράπεζες σε, τέτοιους, σε τέτοιους καιρούς α, είναι άσχημο και πρέπει επίσης να λάβουμε και υπόψη τις επιπτώσεις που έχει στον αποκεντρωμένο τομέα των τραπεζών. Γιατί εμεί πάντα λέγαμε ότι θα πρέπει να δούμε και τον τομέα αυτό. Α μην, τον, ας μην το ξεχάσουμε και ας μην το κρύψουμε κάτω από το χαλί το πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ. Thank you, Udo. Danke, Frau Vorsitzende. Äh, stimme Kollegen Karas zu. Ευχαριστώ. Εγώ συμφωνώ με τον συνάδελφο Κάρας der die wir nicht verstehen. Τα προβλήματα δηλαδή που δεν καταλαβαίνουμε καλά ή δεν τα λύνουμε ή τα διαγράφουμε και τα βγάζουμε από την νομοθεσία. Ε, αυτό μας οδήγησε στην κρίση όμως. Κλείνουμε μονίμως την, ε, την πόρτα και δεν λύνουμε τα προβλήματα και αυτό φυσικά μας οδηγεί σε τελείως αντίθετα αποτελέσματα. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ε, πολύ ε, ενθαρρυντική προσέγγιση που έχει λάβει ως προς το θέμα. Ξέρω ότι έχετε την πλήρη υποστήριξη της ομάδας σας. Η δική μου ομάδα θα ασχολήθηκε κυρίως με το θέμα της μόχλευσης και της επαναδιτλοποίησης και τις αποζημιώσεις, τα μπόνους, ε, ο τρόπος όμως με τον οποίο το αντιμετωπίζετε εσείς, νομίζω ότι θα μπορέσει το Κοινοβούλιο να ε, λάβει τον ρόλο που του αρμόζει. Ε, να, να μπει δηλαδή στη θέση του οδηγού στη σχετική συζήτηση για την του, για τη ρύθμιση συγγνώμη, του τραπεζικού συστήματος. δεν θα χρησιμοποιήσω άλλο χρόνο για να μπορέσουν να προλάβουν και οι υπόλοιποι να μιλήσουν. Και θα ήθελα και εγώ να ζητήσω τις απαντήσεις της Κομισιόν. πραγματικά έχει θέσει πολύ σωστά ερωτήματα η εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να πω στην εισηγήτρια ότι μας υπέβαλε πολλές ερωτήσεις, αλλά ουσιώδεις ερωτήσεις. Αυτή τη στιγμή που μας απασχολούν διάφορα χρηματοπιστωτικά ζητήματα και συμφωνώ με τον Ότμαρ ότι χρειάζεται μια συνοχή μεταξύ των ζητημάτων όσο μας απασχολούν θα πρέπει να υποβάλουμε όλο ένα και περισσότερο πολιτικά ερωτήματα. Δεν θα πρέπει να εμπλακούμε σε τεχνικές συζητήσεις όπου κάτι καταλαβαίνουμε ή τουλάχιστον μερικοί από εμά και να κρυφτούμε πίσω από δέντρα. Όπως ξέρετε, είμαι εισηγητής στο IFM και γνωρίζω, έμαθα ότι έχουν υποβληθεί 1.300 τροπολογίες. Είναι ρεκόρ για την Επίτροπη Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Δεν τις ανέλησα. Ορισμένοι συνάδελφοι μου απέστειλαν τις βασικές τροπολογίες. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτός ο αριθμός των τροπολογιών ε, ε, αφορά ζητήματα ύψης της σημασίας και το πόσο βάζουμε ένα λιθαράκι κι εμείς ή αυτό αφορά μόνο μερικές από αυτές. Μερικές θέλουν να θολώσουν και τον ορίζοντα. Και μερικέ μας λένε δεν καταλαβαίνετε τίποτα έτσι κι αλλιώ σα το διανθίσουμε. Σε αυτό το χρηματοπιστωτικό ζήτημα θα πρέπει να υποβάλουμε σαφείς ερωτήσεις. Πού έγκυται το γενικό οικονομικό συμφέρον της Ευρώπης και των συμπολιτών και γενικότερα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πού έγκυται το συμφέρον της ευρωπαϊκής οικονομίας. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη και την βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και να λάβουμε υπόψη και έρευνες που λαμβάνουν ε, υπόψη ε, το γενικότερο οικονομικό συμφέρον. Εάν χαθούν χίλιες θέσεις κερδοσκόπων, αυτό δεν με δυσαρεστεί ιδιαίτερα. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη την χρηματοπιστωτική βιομηχανία, η οποία πρέπει να χρηματοδοτεί την οικονομία και να δημιουργεί πλούτο και όχι τεχνητό πλούτο με δημιουργικές λογιστικές, επενδύοντας σε πιο αποδοτικούς τομείς και, εν περιπτώσει, δεν θα πρέπει να είναι μία βιομηχανία που να ομφαλοσκοπεί. Αυτό σημαίνει σκέψη, να είμαστε θαραλέοι και να θέλουμε να εξεύρουμε ένα εξισορροπημένο χρηματοπιστωτικό σύστημα, να μην είμαστε ουραγοί αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Ας σκεφτούμε συλλογικά έτσι ώστε η χρηματοπιστωτική ευρωπαϊκή βιομηχανία να είναι αποτελεσματική και να υπηρετεί το γενικό οικονομικό συμφέρον. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Πασκάλ θα ήθελε τώρα να λάβει το λόγο γιατί είναι και σκιώδης. Euh, Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρη για την ποιότητα των ερωτήσεών της. Ιδιαίτερα όταν μας λέει ότι οι τράπεζες ε, θα πρέπει να υπηρετούν την οικονομία χωρίς να χορηγούν αλόγιστα μπόνους τη στιγμή που δεν υπάρχουν ε, σαφείς δεσμεύσεις και δεσμευτικοί κανόνες. Αναφερθήκατε στην φορολόγηση των μπόνους από την Γαλλία όπως ε, και επειδή αναφερθήκατε θα ήθελα να επανέλθω αυτή η φορολόγηση των μπόνους είναι επιπρόσθετα χρήματα. Δηλαδή δεν βγαίνουν από τις τράπεζες. Απλώς αφαιρούνται από την φορολόγηση των πόνους. Δηλαδή δεν φορολογούνται τώρα οι αμοιβέ, φορολογούνται τα πόνους. Όταν κάνουμε μια τελική αποτίμηση λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι προσθέθηκε αλλά και τι αφαιρέθηκε. Διαφορετικά έχουμε πολύ επιμερισμένη ε, αντιμετώπιση του ζητήματος. Τουλάχιστον στη Γαλλία έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν ξέρω τι ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Τμαρ Καράς είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση της ε, ε, ρύθμισης ως προς το ΣΕΡΔΕ 3, 4 και 5 δεν μπορούμε να θέτουμε τροχοπέδι στη νομοθετική διαδικασία, γιατί όπως είπε και ο κύριος Γκοζές, τότε θα χρονοτριβούμε. Δηλαδή, είτε περιμένουμε αποφάσεις από τους άλλους, δηλαδή όταν τις λάβουν τις ενσωματώνουμε, ή προσπαθούμε να αποφανθούμε επί θεμάτων έτσι ώστε να βρούμε τη σωστή, μια σωστή εξισορρόπηση για να δούμε πώς θα ρυθμίσουμε και στο, το ΣΕΡΔΕ 3. Υπάρχει συλλογική πολιτική θέληση έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μην καταγράφει απλώς το ότι αποφασίστηκε στη ναι, Βασιλεία. Ναι, ναι. Υπάρχει το θέμα της τίτλοποίησης που είναι περίπλοκο. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε επί ενός πιο φιλόδοξου σχεδίου από ε, εκείνο της ε, Βασιλείας. Όταν υπάρχει περίπλοκη τυπλοποίηση, τα προϊόντα είναι πιο περίπλοκα, λιγότερο διαφανή, άρα δεν είναι σίγουρη και η αποτελεσματικότητα των αγορών. Αν δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα. Να δούμε δηλαδή πού υπάρχει συλλογικό συμφέρον. Και όταν ε, κάνουμε έναν απολογισμό βλέπουμε πολλές φορές ότι υπάρχουν περισσότερα μειονεκτήματα παρά πλεονεκτήματα. Άρα ας αποστείλουμε ένα μήνυμα πέρα από την τεχνική συμφωνία της Βασιλείας. Και για να επεκταθώ σε αυτά που είπε ο κύριος Γκοζές, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και με τις αμοιβέ. Αυτό συζητήθηκε και στη Βασιλεία αλλά και στους G20. Θα επανέλθουμε βεβαίως, αλλά καταρχήν θα πρέπει να ορίσουμε ένα όριο σε σχέση με το, το μεταβλητό στοιχείο αυτό επί των αμοιβών. Άρα η μεταβλητή αυτή ε, συνιστόσα να αποτιμάται με βάση ένα σχέδιο μπόνους μάλους. και ως προς τα εγγυημένα μπόνους ε, αποτελούν κίνητρο για να αλλάζει κανείς εργασία. Δηλαδή, ανά δύο χρόνια, μάλλον όταν πρώτο διορίζεται κανείς, έχει εγγυημένο μπόνους για δύο χρόνια. Άρα έχει κίνητρο να αλλάζει εργασία. Θα πρέπει να το δούμε και αυτό. Πίτερ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Αρλίν για την εισήγηση Ίσως θα πρέπει να ψυχολογήσουμε και την όλη κατάσταση, διότι έχουμε ε, συμπεριφορικά πρότυπα. Και άρα πολλοί πάνε στον χρηματοπιστωτικό τομέα για τα μπόνους μόνο και μόνο και για τίποτα άλλο. Αυτό θα πρέπει να είναι το επίκεντρο των σκέψεών μας. αλλά ως προς την προσέγγιση του κινδύνου θα πρέπει να το δούμε, διότι το βλέπουμε και σε επίπεδο φερεγγιότητας. Η παρούσα κρίση δείχνει ότι οι τράπεζες έκαναν ό,τι έπρεπε ως προς τις ε, καταβολές και τις πληρωμές. Τώρα, τι έκανε ο Ομπάμα και δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να τον ακολουθήσουμε. Δεν ξέρουμε καταρχήν αν όλα αυτά θα εισακωστούν από το Κογκρέσο. Θα πρέπει να υπάρχει και μία ευρωπαϊκή ανταπάντηση που να ανταποκρίνεται στα παγκόσμια δεδομένα σε ορισμένες χώρες εκτελούν τους τραπεζίτες. Στην Κίνα νομίζω έγινε αυτό τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν θα ήθελα να το φέρω στο προσκήνιο το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομο γιατί όσοι μίλησαν ήδη ανέφεραν τα πιο σημαντικά. Είναι αναφυσβήτητο ότι οι τράπεζες ε, έχουν, χρειάζονται και ποιοτικό και προσωπικό περισσότερο κεφάλαιο. Ε, πρέπει λοιπόν να, διευκρινίσουμε με ποιο, σε ποιο χρόνο μπορούμε να περιμένουμε να, οι τράπεζες να φτάσουν σε αυτό το υψηλότερο κεφάλαιο. Είναι διαφοροποιημένο το ερώτημα αυτό, γιατί έχουν σήμερα κεφάλαιο το οποίο στο μέλλον δεν θα ε, περνά τις εξετάσεις ουσιαστικά. Ε, έχουμε και τους διαφορετικούς συντελεστές. Υπάρχουν νέες προκλήσεις για το ίδιο κεφάλαιο. Θα είναι λοιπόν πραγματικά πολύ απαιτητικό ο χρόνος αυτός και πρέπει σίγουρα να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα εστευλώσουμε την, ε, το level playing field. Να μην έχουμε δηλαδή δεσπόζουσες θέσεις έναντι κάποιων τραπεζών έναντι κάποιων άλλων. Οι ε, τράπεζες πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, να κινητοποιούν την ε, οικονομία και πέρα από τα χρονικά όρια και τα υπόλοιπα, θεωρώ ότι υπάρχει κίνδυνος, όπως και με τη Βασιλεία 1, να μην ε, λειτουργούμε εμείς παράλληλα με τις ΗΠΑ ε, ή ΗΠΑ παράλληλα με εμάς. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει η Αμερική και η Ευρώπη να βρίσκονται σε ένα ε, στρατόπεδο και να μην έχουν δύο διαφορετικές γραμμές. Ένα ερώτημα που θα ήθελα να θέσω σε αυτά που έθεσε και η Αρλίν το ίδιο κεφάλαιο και η πρικοδότηση με ίδιο κεφάλαιο, το κεφάλαιο είναι ένα εργαλείο ώστε να αντιμετωπίσουμε το ότι οι τράπεζες, κάποιες τράπεζες είναι πολύ μεγάλες για να αποτύχουν. Δηλαδή, πρέπει να θέσουμε ένα συγκεκριμένο όριο, επίπεδο ιδίου κεφαλαίου που μπορεί να είναι ας πούμε δυσανάλογο ώστε να μην είναι πλέον ε, ελκυστικό για μια τράπεζα. Σε ό,τι αφορά τις εγώ πρέπει να πω προσωπικά, γιατί πριν έρθω στο κοινοβούλιο ήμουν 38 χρόνια στην, στον τομέα της οικονομίας, θεωρώ ότι δεν, γίνεται, δεν είναι δικό μας θέμα να ρυθμίσουμε τα θέματα των αποζημιώσεων. Δεν μπορούν να ασχολούνται οι πολιτικοί με αυτά. Αλλά αυτή η έλλειψη διαφάνειας που υπάρχει μας αναγκάζει να ασχοληθούμε, μας αναγκάζει να υποχρονόμαστε να λύσουμε το πρόβλημα. Ο πρόεδρος της Goldman, της Goldman από την Γερμανία είπε ότι οι τράπεζες δεν έχουν καμία κοινωνική ευθύνη. Τελικά δεν έχουν καταλάβει καθόλου τι γίνεται και δυστυχώς όταν λένε τέτοια πράγματα μεγάλοι τραπεζίτες πρέπει να επέμβουν οι πολιτικοί. Πρέπει να δούμε και αυτό το θέμα του μπόνους μάλλον, αλλά κάτι είναι απόλυτα φυσιολογικό και το είδα και στον τομέα της βιομηχανίας. Όταν η εταιρεία δεν έχει επιτύχει τον προϋπολογισμό της, ακόμη και αν ο προϋπολογισμός ήταν θετικός, όχι αν ήταν μηδενικός ή αρνητικός, τότε δεν υπήρχε μπόνους ακόμη και στις, στα, τμήματα που είχαν κάνει, είχαν κάνει πολύ καλή δουλειά και είχαν επιτύχει τους στόχους τους. Εκεί δηλαδή που πρέπει ο φορολογούμενος να σώσει τις τράπεζες, δεν υπήρξε κανένα μπόνους. Ακόμη και για αυτούς που έκαναν καλή δουλειά. Δυστυχώς αυτό βέβαια δεν θα μπορέσουμε να το πουλήσουμε στους τραπεζίτες, αλλά οι τραπεζίτες πρέπει να καταλάβουν ένα πράγμα πρέπει, να, τα πράγματα, πρέπει όλα τα μέτρα που θα λαμβάνονται να είναι, ε, να είναι νόμιμα. Και το θέμα δεν είναι απλώς να είναι νόμιμα, είναι να είναι και ηθικά. Okay. Um, thanks. μάλιστα, μάλιστα. Τώρα θα μιλήσω κι εγώ, γιατί κι εγώ είμαι σκιώδης για τους φιλελεύθερους. Έχουν βέβαια υποθεί ήδη πολλά, και νομίζω ότι θα έπρεπε η συγγήτρια να αναρωτηθεί για τον ρόλο που έχει το θέμα της ισότητος των φίλων και στα θέματα που συζητούμε. Διότι η Επιτροπή της Βασιλείας δεν εργάστηκε με τον ίδιο τρόπο που είχε ζητήσει η Ένωση. Θα υπάρξουν λοιπόν ορισμένες αξιολογήσεις ειδικά για την Ένωση και βέβαια τις χρειαζόμαστε πρώτες πριν δούμε αν δεχόμαστε τη συνολική δέσμη ή αν χρειάζεται να θέσουμε άλλες προτεραιότητες. Την προηγούμενη φορά που κάναμε ανταλλαγή απόψεων είχα ήδη πει ότι χρειάζονται προτεραιότητες αλλά δεν είμαι ούτε εγώ έτοιμη να το κάνω. Και άρα πρέπει κάποτε κάτι να κάνουμε. για τις ε, ευρείες αποκαλύψεις τα είχαμε πει. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. για να δούμε αν μπορούμε να δεχτούμε τη συνολική δέσμη όπως είπε ο Οτμαρ Καράς. Τα άλλα τα είπαν οι υπόλοιποι. Για την επανασφάλιση Αφού ήδη έχει διαθετηθεί το θέμα της ασφαλίσεως, δεν είμαι βέβαιη ότι χρειάζονται υψηλότερα πρόστιμα για τα περαιτέρω. Αν τα πράγματα φτάσουν μέχρι του σημείου να είναι τόσο πολύπλοκα ώστε να χρειαστεί το μέτρο αυτό, τότε νομίζω ότι η κατακράτηση δεν θα χρειαστεί. Γιατί εγώ θέλω οι τράπεζές μας να συνεχίσουν να ζουν και όχι να αναγκάζονται να κατακρατούν. Να σκεφτούν μόνες τους πρώτα την ίδια τους την ασφάλεια, χωρίς να χρειάζεται η λήψη εξωτερικών μέτρων που θα ζημιώσουν και τους κοινού επενδυτάς και επενδυτρίας. Δεοδός βέβαια δεν θέλουμε να υπάρχουν παρεμβάσεις, αλλά είναι γνωστό ότι μπορεί να χρειάζονται. Όταν ακούμε ότι θα πληρώσουν όλοι όπως έγινε ήδη διεθνώς, ε, αυτό μοιάζει σαν να πρόκειται για ένα μυστικό καρτέλ και δεν το θέλουμε. τι θα λέγαμε όταν λένε ότι οι τράπεζες ε, στο κάτω-κάτω δουλεύουν για τα λεφτά. Ε, άμα και οι στρατιώτες λέγανε ότι δουλεύουν γιατί είναι αιμοδιψείς, τι θα λέγαμε. Θα λέγαμε. Δεν είναι πράγματα αυτά. Για να δεχτούμε τα μπόνους πρέπει να έχουμε και έναν τρόπο μέτρησης αν έχει κερδίσει ένας οργανισμός πολλά χρήματα σε έναν τομέα όπου είναι πολύ εύκολο να κερδιθούν τα χρήματα, είναι λιγότερης αξίας των πόνους. Αφού θέλουμε λοιπόν κάποιο κριτήριο, μπορούμε να πούμε γιατί να υπάρχει πόνους υψηλότερο από το κόστος του κεφαλαίου για να κερδιθεί το ποσοστό που κερδίθηκε. Αυτό δεν είναι σωστό. Από εκεί θα βασιστώ εγώ. Σε αυτό θα βασιστώ. Έχουν εφευρεθεί βέβαια διάφορα καινοτόμα προϊόντα, πολύ εφευρετικά, αλλά νομίζω ότι το κριτήριο πρέπει πάντοτε να είναι να μην υπάρχει αυτό το υψηλότερο μπόνους από το κέρδος. Αυτά είχα εγώ να πω. Η Κομισιόν όμως έχει ορισμένες ερωτήσεις φαίνεται, τεράστιο κατάλογο. Ή μάλλον οι συνάδελφοι έχουν τεράστιο αριθμό ερωτήσεων προς την Κομισιόν. Αν μπορέσει η Κομισιόν λοιπόν να απαντήσει σύντομα, καλό θα ήταν. Αλλιώ να μας θέλετε τις απαντήσεις ηλεκτρονικώς. Ποιος θα μιλήσει για την Κομισιόν, κάποιος φαντάζομαι μπορεί όμως και κάποια. Α, ναι, η Ρουθ, Μπορεί να μιλήσουν περισσότεροι από ένας από εμά, αλλά θα είμαστε όλοι σύντομοι. Εγώ θα μιλήσω για τα ευρύτερα, διότι πολλοί και η συγγήτρια μίλησαν για τις μεταρρυθμίσεις του Ομπάμα, για αυτά που συμβαίνουν στη ΣΥΠΑ γενικότερα και το ότι πρέπει να, για το ότι πρέπει να δούμε γενικότερα τη δομή των τραπεζικών. Αυτά που συμβαίνουν όμως γενικότερα δεν γίνονται στα πλαίσια του CRD3 και της Βασιλείας και τα πριν και τα λοιπά. Πρέπει να δούμε παραπέρα. Πώς θα αντιμετωπίζουμε γενικότερα τις κρίσεις στο μέλλον. Έχουμε την δήλωση της Επιτροπής για την αντιμετώπιση των κρίσεων. Έχουμε ήδη κάνει καμιά εξινταριά διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους και πρόκειται σύντομα να γράψουμε ένα κείμενο γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να φέρονται οι τράπεζες και πώς να αντιμετωπίζουν πιθανές πιτοχεύσεις. Να βρεθούν δηλαδή μηχανισμοί με τους οποίους ο τομέας να πληρώνει για τις πτωχεύσεις και τις αποτυχίες. Περίπου αυτό λένε και οι προτάσεις του Ομπάμα, αλλά οι δικές μας θα συνεχίσουμε την επεξεργασία τους και φέτος. Και τώρα θα συνεχίσει ο συνάδελφός μου εδώ πίσω. Και εγώ ευχαριστώ. Για να αρχίσω με τη Βασιλεία. Δεν ακολουθούμε απλώς τη Βασιλεία, δεν ισχύει αυτό. Απλώς πήγαμε στη Βασιλεία, ακούσαμε τις συζητήσεις, επηρεαστήκαμε και τους επηρεάσαμε και όλα αυτά για να είναι τα μέτρα αποτελεσματικότερα για την Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη λύση εκτός από την παραγωγή συνεπών κανόνων για όλους. Πράγμα που με οδηγεί στο θέμα της resecuritization που λέμε. Στη Βασιλεία είπαμε ότι Υπάρχουν κανόνες για αυτό που προτείνονται από τη Βασιλεία, από την Επιτροπή της Βασιλείας και θεωρούμε ότι οι κανόνες αυτοί πρέπει να εφαρμοστούν στην Ένωση μέχρι το τέλος του 2010. Βέβαια υπάρχει το ερώτημα του κατοφλίου και των calibration και resecuritization. Θα το λύσουμε και αυτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται η εφαρμογή αυτών των κανόνων εγκαίρως. Μέχρι το τέλος του 2010 το είπα και πριν. Βέβαια η κρίση είναι πολύπλοκη και πρέπει να εξετάσουμε όλες τις, τις πτυχές. Γι' αυτό χρειάζεται χρόνος, αλλά δεν αμφισβητεί αυτό τη δυνατότητα να υπάρξει γρήγορη πρόοδος ως προς την εφαρμογή των κανόνων του Trading Book. Τώρα έρχομαι στο άρθρο, α όχι με συγχωρείτε, αλλά η περιμένει ο υπουργό, οπότε παρακαλώ καταλήξτε εκεί πέρα γιατί έχουμε υπουργό, τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά. Με συγχωρείτε που σας πιέζω, αλλά, αλλά περιμένει ο υπουργό σας, το είπα δύο φορές. Δεν έχω άλλο χρόνο να σας διαθέσω. Κυρία εισηγήτρια, όχι δεν θα απαντήσω σε όλα όσα υπόκεινα αλλά θα ευχαριστήσω τα μέλη που τα έθεσαν. Θα ήθελα όμως να πω στην Κομισιόν ότι δεν συμφωνώ με την πρότασή σας που λέει ότι πήγαμε στη Βασιλεία αλλά δεν ακολουθήσαμε τυφλά αυτά που υπόθηκαν εκεί. Όχι, επηρεαστήκατε αλλά εσείς δεν επηρεάσατε, δεν χρειαζόταν να περιμένετε τη Βασιλεία για να προτείνετε αυτά που προτείνετε. Γιατί τώρα βιάζεστε κιόλα. Δεν είναι σωστός τρόπος αυτός νομοθετήσεως. Και νομίζω ότι γενικά και οι συνάδελφοι διαφωνούν με τη μέθοδο αυτή. Εγώ τουλάχιστον θα προτείνω μία πολύ ισχυρή μεταρρυθμιστική, ρήτρα μεταρρύθμισης που θα προβλέπει αλλαγές των προτάσεων αυτών επί όλων των σημείων που φύγουμε. Και η πρόεδρος είπε ορισμένα από αυτά γιατί το θέμα δεν είναι να πηγαίνουν εκεί οι τραπεζικοί να έχουν υψηλούς μισθούς και να παίρνουν και πρίμα. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουν οι τράπεζες να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους που συμφέρει ολόκληρη την κοινότητα για να υπάρχει δημιουργία θέσεων επεξεργασίας. Η υπερβολική ανάληψη κινδύνου ή η ανάληψη υπερβολικών κινδύνων είναι θέμα των τραπεζών και όχι των υπολείπων. Εμείς προτείνουμε άλλα πράγματα από την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ και εσάς και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Θα συνεχίσουμε άλλη φορά.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 Right. Oops. Okay. Thank you. Thank you, colleagues. Um, and I, I, if we could, if we could settle down. Um. Παρακαλώ, συνάδελφοι, καθίστε. Ζήτησα συγγνώμη από την ε, Υπουργό, διότι είχαμε μία ενθουσιώδη και ζωηρή συζήτηση, είχαμε μία γεμάτη μερίσια διάταξη, θα προβούμε σε ανταλλαγή απόψεων με την ε, Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της Ισπανίας. Θα μας κάνει μια εισήγηση ενός Τετάρτου και μετά θα έχουμε έρωτα ε, αποκρίσεις, μια σειρά αποκρίσεων. Η Υπουργός έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη χαρά για μένα να βρίσκομαι ενώπιον αυτής της Επιτροπής για να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα της Ισπανικής Προεδρίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί τους πολίτες της Ευρώπης και ενισχύθηκε με τη συνθήκη της Λισαβόνας και τη θέση της σε μέσα από μια νέα νομοθετική διαδικασία. Θα ήθελα λοιπόν να συνεργαστούμε στενά έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις σοβαρές προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Όπως γνωρίζετε, είχαμε προβλέψει μια συνάντηση στα πλαίσια της Τρόικα στις 15 Φεβρουαρίου πριν από το Eurogroup. Κατανοώ βεβαίως ότι εκείνη την εβδομάδα θα ασχοληθείτε με την εργασία στις εκλογικές σας περιφέρειες. La Και έτσι θα βρεθούμε το Μάρτιο. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με βάση τα αποτελέσματα της Σουηδικής Προεδρίας. Ελπίζουμε να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία όπως είχαμε μέχρι τώρα και με το Βέλγιο και με την Ουγγαρία πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και συντονισμό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Κομισιόν και το Συμβούλιο και κυρίως με εσά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι 18 επόμενοι μήνες είναι ζωτική σημασίας έτσι ώστε να υπάρξει ένας βιώσιμος ρυθμός ανάπτυξης. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές αδυναμίες των κυβερνήσεών μας, προωθώντας ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος που αντιμετωπίσουμε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να σταθούμε στην ανάγκη βελτίωσης του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ολοκληρώσουμε την εσωτερική αγορά και για να έχουμε ένα level playing field για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νέα θεσμική αρχιτεκτονική συμπίπτει με την ανάληψη της Ισπανικής Προεδρίας. Και αυτό σημαίνει μια νέα φάση στην οικοδόμηση της Ευρώπης. Όπως γνωρίζετε, η Ισπανική Προεδρία συμπίπτει με το νέο Διευθυντήριο των Επιτρόπων, το διορισμό των Επιτρόπων. Όλα αυτά έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ατζέντα πρωτοβουλειών της Κομισιόν. Η Προεδρία είναι έτοιμη για να ανταποκριθεί στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να φτάσει στις σωστές συμφωνίες με το Συμβούλιο για να ολοκληρώσουμε ή να προωθήσουμε τουλάχιστον αυτή την οικοδόμηση. Θα ήθελα να σας σκιαγραφίσω τις προτεραιότητές μας κατά το επόμενο εξάμεινο. Προτεραιότητες που έχουν ως στόχο την οικονομική ανάκαμψη έτσι ώστε να μην ζήσουμε άλλη κρίση, χρηματοπιστωτική κρίση παρόμοιας εμβέλειας. Αυτό που έχει σημασία είναι να ξεπεράσουμε τη μεγάλη κρίση και να ενδυναμώσουμε, να ενισχύσουμε την, τον πλούτο μας και την ευημερία μας. Η Ευρώπη χτίστηκε πάνω στην κρίση της, στην αρχική κρίση της ύπαρξης της Ευρώπης. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις με βάση συγκεκριμένες πραγματώσεις. Εμείς είμαστε ευρωπαϊστές. Θα υπερβούμε τις δυσχέρειες και θα αφήσουμε το αποτύπωμά μας και εμείς. Προβάλλουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα εργασίας, γι' αυτό θα επικεντρωθώ στα βασικά στοιχεία της δραστηριότητάς μας κατά τους επόμενους μήνες. Σε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά πλαίσια, η πλαισίωση, βρισκόμαστε σε μία στιγμή όπου διαπιστώνουμε την απαρχή μιας ανάκαμψης του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Θα πρέπει να φτάσουμε σε μια βιώσιμη στρατηγική ανάκαμψης και υπέρβασης του κινδύνου για να δούμε τι φορολογικά μέτρα θα προβάλλουμε, έκτακτα φορολογικά μέτρα και έναν βιώσιμο ρυθμό ανάκαμψης. Κατά την Σουηδική Προεδρία ορίστηκαν αρχές που εμείς υλοποιούμε και πραγματώνουμε με τη σειρά μας, έτσι ώστε να προβάλλουμε μια βιωσιμότητα στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό πλαίσιο. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να ορίσουμε χρηματοπιστωτικά ορόσημα για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των χρηματοπιστωτικών αγορών. Πρόκειται για χρηματοπιστωτικά συστήματα τα οποία βρίσκονται σε μια μεταβατική φάση και θα φτάσουν σε μια αυτονομία χωρίς την στήριξη των κυβερνήσεων. Σε σχέση με τα δημόσια οικονομικά, πιστεύω ότι το στοιχείο κλειδί είναι το σύμφωνο σταθερότητας. Θα πρέπει να δράσουμε με αυστηρότητα έτσι ώστε να μειώσουμε τα ελλείμματα εν ευθέτω χρόνο. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε όμως να κινηθούμε πέρα από την μείωση των ελλημάτων, των δημοσίων ελλειμμάτων. Θα πρέπει να φτάσουμε σε μία χρηματοπιστωτική ανάκαμψη για να έχουμε μακροχρόνια βιωσιμότητα. Αυτή τη στιγμή 20 από τα 27 κράτη-μέλη έχουν ε, ανοιχτές διαδικασίες εξαιτίας υψηλών ελλημάτων. Στο επόμενο και στα επόμενα εκοφήν θα δούμε κατά πόσο τα κράτη αυτά μπόρεσαν να διορθώσουν τα υπερβολικά ελλείμματα με βάση τους στόχους του ΕΚΟΦΗΝ του παρελθόντος Ιουλίου. Αυτό αφορά ιδιαίτερα την Ελλάδα, διότι θα, μπορούσαν, θα να υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις για το ευρώ και την εμπιστοσύνη των χρηματοπιστωτικών αγορών. Άρα θα επικεντρωθούμε όχι μόνο στην απόσυρση των, της δημόσιας στήριξης, αλλά θα ασχοληθούμε και με μια αρχιτεκτονική εποπτείας. Το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο θα ασχοληθεί με αντιμετώπιση ζητημάτων συστημικού κινδύνου και θα συμφωνήσουμε ως προς την οδηγία Omnibus 1 μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την πρόταση οδηγίας Omnibus 2 εάν υποβληθεί κατά την Προεδρία μας. Η χρηματοπιστωτική διασφάλιση είναι ύψης της σημασίας με βάση τα όσα όρισε το ΕΚΟΦΗΝ τον παρελθόντα Ιούνιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τον ίδιο μήνα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο έφτασε σε μια γενική συμφωνία ως προς το, ως προς το σχέδιο μικροεποπτείας που είχε προταθεί ήδη τον Οκτώβριο. Έχουμε λοιπόν δύο σχέδια. Τον Οκτώβριο μικροεποπτεία, σχέδιο μικροεποπτείας και μακροεποπτείας. Οκτώβριο και Δεκέμβριο αντίστοιχα. Έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το όλο χρηματοπιστωτικό πλαίσιο ανάπτυξης όπως ορίστηκε τον Ιούνιο από το ΕΚΟΦΗ. το Συμβούλιο θα συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να φτάσουμε σε μία συμφωνία χωρίς ε, καθυστερήσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο, με βάση αυτή τη νέα αρχιτεκτονική χρηματοπιστωτικής εποπτείας, θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, να προωθήσουμε αυτά τα μέτρα ήδη κατά το τρέχον έτος. Θα πρέπει να δώσουμε μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μία διαδικαστική πορεία, γιατί για πρώτη φορά τίθεται ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο σε σχέση με όλα τα ταμεία επενδύσεων. Όπως όρισαν και οι G20, το Συμβούλιο εργάστηκε σκληρά επί των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε να φτάσουμε σε μια νέα νομοθετική συμφωνία κατά τις επόμενες εβδομάδες για ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο και εξετάσαμε τις ε, προτάσεις του κυρίου Γκοζές που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση με αυτήν του Συμβουλίου. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα επιτύχουμε μια συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωρίς δυσχέρειες. Το optimum θα ήταν να φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση. Συνεχίζονται οι εργασίες και σε άλλες προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου που βρίσκονται επιτάπητος. Πιστεύουμε ότι θα αρχίσουμε με τις ε, διαπραγματεύσεις ως προς ε, την οδηγία ρύθμισης της κεφαλαιαγοράς. Το κείμενο αυτό θα επικαιροποιηθεί για να λάβουμε υπόψη τις αλλαγές μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας πριν αρχίσουμε τις διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο. Σε σχέση με την οικονομική στρατηγική για το μέλλον, κατά τους επόμενους μήνες θα κινήσουμε, θα κινήσουμε την διαδικασία, την ε, πρότασή μας Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος. Θα πρέπει λοιπόν να ορίσουμε όχι μόνο τους κατάλληλους στόχους, αλλά και τα μέσα τα οποία επιβάλλονται για την επίτευξη των στόχων αυτών. Αυτό είναι ένα κεντρικό σημείο της ευρωπαϊκής μας πολιτικής και η Ισπανική Προεδρία έχει δεσμευτεί έτσι ώστε να ευεργετηθούμε από αυτή τη νέα στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 και αυτό μέσω πρόθεσμα. Όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 11 Φεβρουαρίου θα συνέλθει για να δώσει ορισμένες αρχικές κατευθυντήριες γραμμές για τις μελλοντικές μας εργασίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεισφέρει και εκείνη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το ΕΚΟΦΗΝ θα πρέπει να συνεισφέρει άμεσα mm. για να εξασφαλίσουμε μια επιτυχή στρατηγική και να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και των προκλήσεων. Δεν είναι εύκολο αυτό το καθήκον. Θα πρέπει να λάβουμε δύσκολες αποφάσεις, όμως θα πρέπει να προωθήσουμε μια συντονισμένη και συνεκτική στρατηγική. Η Ισπανική Προεδρία θα αξιολογήσει αυτές τις εργασίες για να φτάσουμε στον επιδιωκόμενο στόχο. Ε. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο στα πλαίσια της παγκόσμιας οικονομικής συνεργασίας, ιδιαίτερα σε επίπεδο G20, που μετατρέπεται σε βασικό φόρουμ, παγκόσμιο φόρουμ επί οικονομικών θεμάτων. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις με βάση εύρωστες και στεναρές θέσεις, τόσο σε επίπεδο υπουργών οικονομικών και διοικητών κεντρικών τραπεζών. Επίσης, οι χρηματοπιστωτικές αρχές παγκοσμίως μεταρρυθμίζονται. Θα πρέπει να υπάρχει μια ευρωπαϊκή εποπτεία και ένα ευρωπαϊκό όραμα έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις για το μέλλον των χρηματοπιστωτικών παγκοσμίων οργάνων. Κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας θα ασχοληθούμε με το ρόλο της ΕΤΕ, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη το ρόλο των αναδυόμενων οικονομιών όπως της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. Mm. Θα προωθήσουμε και τη διεθνή οικονομική συνεργασία, ιδιαίτερα στα πλαίσια των χωρών της ε, Μεσογειακής Λεκάνης. Τέλος, σε σχέση με το φορολογικό πλαίσιο, θα προωθήσουμε την διαφάνεια και ένα πλέον αποδοτικό φορολογικό σύστημα το οποίο να προβάλλει πιο στενή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ε, φοροδιαφυγή. Αυτό αφορά άμεση και έμεση φορολόγηση. Θα βασιστούμε στις τρεις προτάσεις οδηγίας για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και συναφών παρεπόμενων μέτρων. Επίσης, θα προβούμε σε ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες. Στο ΕΚΟΦΗΝ της προηγούμενης εβδομάδας φτάσαμε σε μία συμφωνία γενικών κατευθυντήριων γραμμών ως προς μία πολιτική εισφορών και εισπράξεων, φοροεισπράξεων. Η οδηγία αυτή είναι η πρώτη που ενεκρίθη μέσα στα πλαίσια ενός πακέτου χρηστής οικονομικής διακυβέρνησης. Θα προωθήσουμε και τα παρεπόμενα διοικητικά μέτρα. Ξέρετε ότι χρειάζεται ομοφωνία για αυτές τις προτάσεις. Προωθήσαμε έναν επικοδομητικό διάλογο, έτσι ώστε να αναζητήσουμε λύσεις συμβιβασμού που να γίνονται αποδεκτές από όλους. Η Ελλάδα, η, η Προεδρία με συγχωρείτε, θα συνεργαστεί διμερώς με τις χώρες που επιβάλλεται και θα προωθήσουμε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου να προωθήσουμε αυτές τις προτάσεις οδηγίας. Επίσης, στα πλαίσια της ε, φορολογίας θα ασχοληθούμε με θέματα εσωτερικής αγοράς θα ασχοληθούμε με τον ΦΠΑ mm. και άλλες ε, έμεσες μορφές φορολόγησης. Στα πλαίσια του ΦΠΑ θα προωθήσουμε το Eurofisc έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την απάτη, τη φορολογική απάτη διακοινωτικά και να ορίσουμε ενιαίους κανόνες τιμολόγησης. Θέλουμε να υπάρχει ένα καλύτερο και πιο αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα ιδιαίτερα σε σχέση με τη φορολόγηση υπέρ του περιβάλλοντος. Αυτό θα βοηθήσει και τον ενεργειακό τομέα και την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Γι' αυτό καλωσορίζουμε την πρόταση τροποποίησης της οδηγίας για την φορολόγηση προϊόντων ενεργείας και θα την εξετάσουμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Επίσης, θα ασχοληθούμε και με μία άλλη πρωτοβουλία. Να μειώσουμε τη γραφειοκρατία που βαρύνει τις επιχειρήσεις μέσω της ε, φορολόγησης, μάλλον της ε, ηλεκτρονικής φορολόγησης για τον ΦΠΑ, του ΦΠΑ. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο και ελπίζω να τα καταφέρουμε με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να φτάσουμε στους ε, στόχους τους οποίους επιδιώκουμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων για τις ερωτήσεις σας και είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ. Um, ευχαριστώ. Όντως είναι γεμάτη η ατζέντα σας. Και εμείς ε, ε, εξίσου πολλή δουλειά έχουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις μαζί σας για διάφορα θέματα από αυτά που ήδη θίξατε. Ben Giegold, Udo Bullman, Pablo Zalva Bidigan, uh, Annika Gyuri and Antolin Sanchez Presedo. Uh, I've now got, hang on, Tremosa, Alvarez. Anybody else? Was was that? No, no, no. Right. Oh, uh, and Theo. Okay, right. Well, we'll make a start. So first. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Να ακούσουμε τον Αντιπρόεδρο καταρχήν. Ευχαριστώ να καλωσορίσω και εγώ την Αντιπρόεδρο με τη σειρά μου. Το θέμα της χρηματοπιστωτικής εποπτείας είναι ύψης της σημασίας. Είναι το πιο δύσκολο θέμα που αφορά τις διατραπεζικές ή διασυνοριακές συναλλαγές. Πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ένα διασυνοριακό εποπτικό σύστημα. Αυτό που έχει σημασία, λοιπόν, είναι να ζητήσουμε τη συνεργασία των εθνικών εποπτικών αρχών, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην κρίση. Η συμφωνία σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προτείνει το ίδιο, δηλαδή καλύτερη εποπτεία και σε εθνικό και σε υπερεθνικό επίπεδο. Θα πρέπει όμως όπως υπενθύμησαν οι τέσσερις ε, μεγάλες πολιτικές ομάδες, να επιτευχθεί μια πιο διευρυμένη συμφωνία, η οποία δεν επετεύχθη επί Σουηδικής Προεδρίας. Κάτι το οποίο είναι απολύτως αναγκαίο για μια διασυνοριακή εποπτεία. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη και περισσότερη εποπτεία κατά συνέπεια για να δώσουμε μία σαφή απάντηση. Τι πιστεύετε ως προς την διασυνοριακή εποπτεία για να αντιμετωπίσουμε τους ε, συστημικούς κινδύνους. Θα πρέπει να υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Αρχή Διασυνοριακής Εποπτείας, η οποία να μπορεί να δρά με τη συνεργασία των ε, εθνικών εποπτικών αρχών, που θα ακολουθούν οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Αρχή. Έτσι αποφεύγουμε γραφειοκρατία και ισχύουν τα ίδια κριτήρια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα είχαμε την σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου που θα συγχρηματοδοτήσουν εθνικές ιδιωτικές αρχές όπως ισχύει στην περίπτωση της Ισπανίας για τα κεφάλαια, για την εγκυοδοσία κεφαλαίων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις αρχές ή τους φορείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και για να μην ε, επομιστούν το κόστος οι φορολογούμενοι, όπως ε, ανακοίνωσε και ο πρόεδρος Ομπάμα. Εάν ε, λοιπόν επικρατήσει μια ευρωπαϊστική τάση, τότε θα μας ακολουθήσετε σε αυτό το ταξίδι που θέλουμε να ξεκινήσουμε. Έτσι ώστε τουλάχιστον να, υπάρχουν, να υπάρχει ένα ελάχιστο κατόφλι το οποίο θα μπορέσουμε να δεχτούμε σε ευρωπαϊκό ε, επίπεδο σε σχέση με, τις, ε, με μια Ευρωπαϊκή Αρχή Διασυνοριακής Εποπτείας. Επειδή είσαστε οι δύο επόμενοι ομιλητές είναι εισηγητές σε σχέση με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, θα ήταν σκόπιμο να συμπτύξετε τις ερωτήσεις σας. Όταν ε, κανείς... Ξέρετε ότι συνήθως οι κοινοβουλευτικοί ρωτάνε πολλές ερωτήσεις και δεν γνωρίζετε την απάντηση, αλλά Γι' αυτό θα σας συγχωρήσουμε, δεν έχουμε πολλές απαιτήσει. Απλώς νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει κάτι σύντομα για την εποπτεία. Και υπάρχουν τρεις εισηγητές, εγώ, ο Γκαρσία Μαργκάλιου και άλλους, που έχουμε γράψει επιστολές όπου σας ζητάμε βοήθεια, ιδιαίτερα για το θέμα της φορολογικής ευθύνη, που είναι ένας από τους τομείς που είναι οι λεπτότεροι. Και για χρειαζόμαστε απαντήσεις σαφέστερες από την Προεδρία και αν δεν μπορείτε σήμερα κάποια συζήτηση πρέπει να γίνει. Δεν θέλουμε να υπάρχουν καταχρήσεις των όρων που χρησιμοποιούνται. Ξέρω ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο, αλλά το Κοινοβούλιο θέλει να επιμείνει και χρειάζεται απαντήσεις. Οι τρεις αυτές εκθέσεις, αν γραφτούν σωστά μπορούν να έχουν πολύ θετικές επιπτώσεις και χρειάζεται επαναλαμβάνω η βοήθειά σας διότι και εμείς θέλουμε να τα πούμε σοβαρά. Γι' αυτό θέλουμε και σοβαρές απαντήσεις. Καταρχάς σας καλωσορίζω και από την πλευρά μας κυρία Υπουργέ μου. Προσβλέπουμε με μεγάλες ελπίδες στην Ισπανική Προεδρία, ιδιαίτερα για την δημοσιονομική εποπτεία, όπου μπορούμε να πάρουμε μαθήματα από σας. Είχατε προβλήματα στην οικονομία σας και ορισμένα τα λύσατε, τουλάχιστον τα τραπεζικά, πολύ καλύτερα από τη δική μου χώρα και μερικές ακόμα που αντιπροσωπεύονται εδώ στην Επιτροπή μας. Παρ' αυτά, όταν φτάσουμε στα διαμεθοριακά θέματα, εκεί έχουμε ορισμένα ερωτήματα και χρειαζόμαστε μεγαλύτερη συνέπεια να επιδείξει η Ένωση γι' αυτό. Δεν μπορώ παρά να υποστηρίξω τις ερωτήσεις που έθιξε ο συνάδελφος Μαγκάλιο. Πώς θα διασφαλίσουμε κάποια διευθέτηση και εποπτεία διενοσιακών των τραπεζικών δραστηριοτήτων με τρόπο που να αποφεύγει τη δημιουργία προβλημάτων που θα τεθούν και στην επόμενη κρίση για την εδαφική ή περιφερειακή δικαιοδοσία. Αυτά που είπε ο πρόεδρος Απατέρο για την οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη και γενικότερα στην Ευρώπη είναι σημαντικά γιατί διαπιστώνουμε μεγάλες ανισότητες στην Ευρωζώνη που επηρεάζουν και τη δική σας και τη δική μου χώρα. Θα θέλαμε λοιπόν να μάθουμε με ποια συγκεκριμένα μέτρα και σε ποιους τομείς θα θέλατε να υπάρξει ενδυνάμωση για ισχυρότερη οικονομική συνεργασία και συντονισμό ώστε να μειωθούν οι ανισότητες αυτές που αποτελούν κίνδυνο για την ακαιρεότητα της εσωτερικής αγοράς. Πώς θα τις περιορίσετε με τι συγκεκριμένα μέτρα. Αν θέλετε κυρία Υπουργέ, για τα θέματα αυτά της εποπτείας και της διακυβέρνησης, σε τρία-τέσσερα λεπτάκια όμως παρακαλώ. Sí, eh. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω μάλλον να σας ευχαριστήσω για τις ερωτήσεις, διότι δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον από τη δική σας πλευρά και τη σοβαρότητα του ζητήματος. Γνωρίζετε ότι αυτή η γενική προσέγγιση, general approach του ECOFIN ελήφθη ομόφωνα. Άρα προσδίδουμε μεγάλη σημασία σε αυτή την ομοφωνία σε επίπεδο ΕΚΟΦΗΝ και είναι υποχρέωσή μου στα πλαίσια της Προεδρίας να πω ότι η Γενική Συμφωνία του Συμβουλίου μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω θετικά βήματα όπως αποφάνθηκε και το ΕΚΟΦΗΝ. Οι εποπτικές αρχές όμως θα πρέπει να αρχίσουν με τις εργασίες τους το συντομότερο δυνατόν θα διαπραγματευτώ, θα συζητήσω, θα προωθήσω αυτό το διάλογο με το Κοινοβούλιο σε συγκεκριμένη βάση. Εμείς προσδίδουμε μεγάλη σημασία στη δράση της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής, των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μειώνεται ο ρόλος των εθνικών εποπτικών αρχών με βάση τις συμφωνίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δηλαδή, οι εθνικές εποπτικές αρχές θα ανταποκριθούν και εκείνες σε αυτό το κοινό έργο για να φτάσουμε σε μια νέα εξισορρόπηση του συστήματος σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο, στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Μαργάλιο και με βάση και τις ε, δηλώσεις του Προέδρου του κυρίου Ομπάμα, ε, θα πρέπει να τονίσω ότι βρισκόμαστε εκτός εποπτικών αρχών και στο άτυπο Συμβούλιο του Απριλίου, στο ΕΚΟΦΗΝ, άτυπο ΕΚΟΦΗΝ του Απριλίου, σε επίπεδο διοικητών κεντρικών τραπεζών θα συζητήσουμε και αυτή και για άλλες προτάσεις που υπάρχουν επιτάπητος πολλές προτάσεις προέρχονται από κράτη-μέλη. Στο προηγούμενο ΕΚΟΦΗΝ η Σουηδία προέβαλε μια συγκεκριμένη πρόταση και άλλες είναι απότοκες προτάσεων των ε, G20. Θα έχουμε λοιπόν μία κάλυψη, μία συνυπευθυνότητα ως προς την κάλυψη κινδύνων με βάση τη συνεργασία ευρωπαϊκών και εθνικών εποπτικών αρχών, όπως είπε και ο Ευρωβουλευτής. Και, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να προβάλλουμε μία συντονισμένη δραστηριότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιμένω όμως ότι πρόκειται κάτι ξεχωριστό πέρα από το πακέτο εποπτείας σε σχέση με τα φορολογικά μέτρα. Ε, κατανοώ την ανησυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα φορολογικά αυτά μέτρα. Στο ΕΚΟΦΗΝ το Δεκέμβριο φτάσαμε στη συμπλήρωση γενικών κατευθυντηρίων γραμμών και κατά τις διαπραγματεύσεις θα δώσουμε μεγάλη ακρίβεια στην ενιολογική αυτή βάση στις προτάσεις κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από τους ορισμούς του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου του 2009. Γιατί τότε μιλήσαμε για μια φορολογική βάση και επιπρόσθετα φορολογικά μέτρα, τα οποία θα οριοθετήσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς τη συνεργασία για την κατάρτιση οικονομικών πολιτικών θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όπως το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, έτσι και εδώ γνωρίζουμε ότι η φορολογική πολιτική μιας χώρας σχετίζεται άμεσα με το δημόσιο χρέος και με το έλλειμμά της. Υπάρχει αιτιώδη συνάφεια και γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ως βασικό όργανο, διότι το οποιοδήποτε έλλειμμα πλήττει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό η στρατηγική 2020 αφορά μεσοπρόθεσμους στόχους και θα δούμε πώς θα ορίσει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτή τη νέα διακυβέρνηση, οικονομική διακυβέρνηση με συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέτρα. Um, Ωραία. Να δούμε τους επόμενους τρεις. Ούντο, Πάμπλο και Ανίκα ύστερα. Frau Ministerin, Καλώς ήρθατε κυρία Υπουργέ. Χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ. Έχω μία παρατήρηση ουσιώδη να κάνω. Καλώς ήρθατε, εξ ονόματος των σοσιαλιστών. Σας καλωσορίζουμε, κύριε Υπουργέ. Έχω μια βασική παρατήρηση να κάνω για το θέμα της νομοθεσίας. Η Επιτροπή μας προσπαθεί να ε, εφαρμόσει να, γρήγορα μια αποτελεσματική νομοθεσία. Θα είμαστε καλοί συνομιλητές μαζί σα Φροντίζουμε γρήγορα να δρούμε. Δεν θέλουμε απλώς να γίνει να υπάρξει μια, α, συν, μια συμφωνία επί της οποίας μετά να πρέπει εμείς εκ των υστέρων να αναγκαστούμε να συμφωνήσουμε. Θέλουμε ενεργά να δράσουμε ώστε επί τη βάση του διαλόγου να έχουμε καλή και αγαστή συνεργασία. Τώρα, για το θέμα της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020 και το τι γίνεται με την ε, χρηματοπιστωτική κρίση και τις επιπτώσεις στην οικονομία και την ε, απασχόληση. Ε, πριν από 10 χρόνια ξεκίνησε να εκπονείται η στρατηγική της Λισαβόνας. Τότε η Κομισιόν είχε πει ότι ε, θα πηγαίνουμε από επιτυχία σε επιτυχία. Παρόλο που τα κράτη-μέλη δεν ήταν και πολυθετικά. Φτάνουμε στο 2010, 2009. Ε, Μετά από 9 χρόνια η Κομισιόν του Μπαρόζο δίνει άλλα, βγάζει άλλα συμπεράσματα και τώρα λέει ότι θα χρησιμοποιήσει νέα στρατηγική. Μας είπαν τελικά ότι δεν πήγαμε από επιτυχία σε επιτυχία τελικά ήταν πλήρη αποτυχία γιατί ακριβώς τα κράτη-μέλη δεν συνεργάστηκαν. Και η Κομισιόν του Μπαρόζο υποβάλλει ένα έγγραφο όπου λέει ακριβώς το ίδιο. Αυτό δηλαδή που υπήρχε πάντα στα διάφορα έγγραφα, με εξαίρεση αυτών που, που αφορούσαν την απασχόληση και την οικονομία. Εγώ θα σας ενθαρρύνω να είσαστε πολύ συνεπείς όταν ε, λέτε ότι μόνο με ε, δεσμευτική πολιτική μπορούμε να προχωρήσουμε. Εσείς πολύ σωστά είπατε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα που πρέπει να λυθούν. Βρήκατε ποια είναι τα κενά. Τα κράτη-μέλη πρέπει να ε, συνεργαστούν. Το πακέτο σταθερότητας και ανάπτυξης είναι σημαντικό. Και πρέπει όλα αυτά να είναι δεσμευτικά για την οικονομική πολιτική. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Μόνο έτσι μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Α είμαστε λοιπόν θαραλέοι και α μην αφήσουμε να παρασυρθούμε από αδιαφωνίε των κρατών μελών. Um, Pablo it's ε, Ευχαριστούμε, κύριε Αντιπρόεδρε. Φέρετε μεγάλη ευθύνη και αντιμετωπίζετε μια μεγάλη πρόκληση. Θα πρέπει να ορίσετε τις βάσεις της μελλοντικής στρατηγικής 2020. Άκουσα με προσοχή τις προτάσεις σας Όπως είπατε, η χρηματοπιστωτική κρίση σημαίνει ότι θα πρέπει να συντονίσουμε καλύτερα τις οικονομικές μας πολιτικές. Επίσης, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι επιλογές που δεχτήκαμε μέχρι τώρα και οι οποίες δεν ήταν αποδοτικές. Άρα η στρατηγική 2020 θα πρέπει να ορίσει νέες εναλλακτικές και υποχρεώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ασχοληθεί με θέματα οικονομικής διακυβέρνησης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς ε, ορίζεται μια οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 27 κράτη-μέλη. Είπατε ότι αναμένουμε μία απάντηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πώς θα λάβετε υπόψη όμως την εκτέλεση και την εποπτεία αυτού του πλαισίου, πώς θα δράσει η Επιτροπή, Συμβούλιο και κράτη-μέλη και πώς τα κράτη-μέλη μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές αυτές προκλήσεις. Μπορεί να υπάρχει μέθοδος ανοιχτού συντονισμού. Χρειάζεται benchmarking. Θα πρέπει να υπάρχει ήπια προσέγγιση Επίσης, μιλήσαμε για τις υπερεθνικές εποπτικές αρχές. Αν καταρακωθεί το οικονομικό σύστημα, ποιος θα φέρει την ευθύνη στα πλαίσια της γενικότερης αυτής εποπτείας. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ. Ε, ως Ευρωβουλευτής από την Ουγγαρία θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Θα συνεργαστούμε στα πλαίσια της Τρόικας και χάρηκα διότι είχαμε την ε, δυνατότητα να συνεργαστούμε και μέχρι τούδε. Έχει συμβολική σημασία το ότι συνεργάζονται μια μεσογειακή χώρα, μια χώρα από τις ιδρυτικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια χώρα της κεντρικής Ευρώπης. Θα συνεργαστούμε για να φτάσουμε στους ε, νέους αυτούς στόχους. Θα συνεχίσω στα αγγλικά. Δυστυχώς δεν μπορώ να μιλήσω την γλώσσα μου σήμερα. Ε, αντίκειται λίγο στα θεμελιώδη δικαιώματα που έχουν οι ευρωβουλευτές, αλλά... Εν πάση περιπτώσει, για αυτή τη στρατηγική λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Κατά τύχη είναι το δικό μου το ερώτημα, σχετίζεται το δικό μου το ερώτημα με αυτό. Είναι πραγματικά μια πολιτική υψηλής προτεραιότητας για τη δική μας Επιτροπή και φαντάζομαι και για όλους τους πολίτες της Ευρώπης, γιατί οι πολίτες μας χρειάζονται θέσεις εργασίας. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι το εξής. Πώς θα μοιραστείτε το άκθος με τον ε, πρόεδρο Φαν Ρόμποϊ. Ε, πώς θα συνεργαστείτε για τη στρατηγική και για την ε, εφαρμογή της. Οι ιδέε σα ποιε είναι, όπω είπαν και οι συνάδελφοι, πώ μπορεί να υπάρχει συνυπευθυνότητα μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων για την εφαρμογή αυτή τη νέα στρατηγική, Γιατί θα είναι πιο αξιόπιστη αυτή η νέα στρατηγική από την αρχική στρατηγική τη Λισαβόνα, πώς θα την εναρμονίσετε με, την υπάρχουσα, με τις υπάρχουσες μάλλον πολιτικές της Ευρώπης, όπως πολιτική συνοχή, σε διαφορετικά ταμεία. Αν μπορούσατε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες ως προς αυτά, ξέρετε το Κοινοβούλιο πραγματικά θέλει να καταλήξει σε κάτι για αυτό το πρόγραμμα. Θα ήθελα λοιπόν να είναι σαφής ο ρόλος του. Ξέρετε ότι μέχρι το τέλος της Προεδρίας σας πρέπει το πρόγραμμα αυτό να είναι ε, να έχει εγκριθεί. Ε, δεν ξέρουμε ποιο ακριβώς θα είναι ο δικό μας ρόλος σε όλη αυτή τη διαδικασία, οπότε αν θέλετε να μας απαντήσετε, πραγματικά θα το εκτιμούσαμε. Ευχαριστώ. Sí, muchas gracias. Ε, Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω και στα τρία ερωτήματα. Δεν υπάρχει επίσημη πρόταση στρατηγικής Ευρωπαϊκή Ένωση 2020. Γίνεται δημόσια διαβούλευση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν απαντήσεις και ανταπαντήσεις, αλλά δεν έχουμε μία επίσημη στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 με αυτή τον τίτλο. Δεν υπάρχει έγγραφο, έτοιμο έγγραφο για το Συμβούλιο της 11 η Φεβρουαρίου. Θα είναι μια ανοιχτή συζήτηση, θα προωθηθεί μια ανοιχτή συζήτηση χωρίς να βασιστούμε σε ένα γραπτό κείμενο. Δεν μπορώ λοιπόν να σας μιλήσω για μια γενικότερη οικονομική διακυβέρνηση. Δεν είναι κάτι εύκολο. Αυτό δεν μπορεί να το ορίσει η Προεδρία. Θα πρέπει να ορίσουμε και να εντάξουμε την οικονομική διακυβέρνηση στη στρατηγική 2020. Ξέρετε ότι το ΕΚΟΦΗΝ διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο για το περιεχόμενο αυτής της στρατηγικής και νομίζω ότι στο εγγύς μέλλον θα μπορέσουμε να δώσουμε την απαρχή μιας απάντησης. θα πρέπει να πρόκειται για μια βιώσιμη στρατηγική απλής περιβαλλοντικής και οικονομικής πλευράς. Άρα το έγγραφο αυτό θα πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτές τις τρεις προαπαιτήσεις. Ρωτήθηκα το κατά πόσο η στρατηγική της Λισαβόνας ήταν μια επιτυχή στρατηγική ή κατά πόσο αμφισβητείται. Θα μπορούσα να προβάλλω μια προσωπική άποψη. Η στρατηγική της Λισαβόνας γνώρισε μεγάλες επιτυχίες, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένους τομείς. τώρα ακούγονται ορισμένα ερωτηματικά σε σχέση με την, ε, τα πλαίσια της διακυβέρνησης που εντάσσεται στη στρατηγική της Λισαβόνας. Στα πλαίσια μιας νέας στρατηγικής 2020 θα ορίσουμε μια μορφή διακυβέρνησης έτσι ώστε 10 χρόνια μετά να μην πούμε ότι απέτυχε η στρατηγική αυτή. Δηλαδή η διακυβέρνηση εντάσσεται, θα ενταχθεί σε αυτή τη στρατηγική 2020 για να υπάρχει συντονισμός επιμέρους οικονομικών πολιτικών. Βεβαίως αυτό μπορεί να γίνει υπό διάφορες μορφές. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα έχουμε έναν ήπιο συντονισμό ή θα προβάλλουμε πιο αυστηρές προαπαιτήσεις. Γνωρίζετε ότι όταν μιλάμε για ήπιο συντονισμό, για συντονισμό soft, αυτός ο συντονισμός δεν είναι αρκετά επαρκής. Όταν μιλάμε για benchmarking ή για peer review, έχει μεγάλη σημασία να δούμε τι εμπλέκεται σε αυτό τον ορίζοντα. Ίσως πρόκειται για μια ήπια προσέγγιση. Εν πάση περιπτώσει ήταν δεσμευτική αυτή η στόχη. Ένα άλλο ζήτημα είναι πώς θα επιτύχουμε αυτούς τους στόχους ή κατά πόσο δεν μπορούν να επιτευχθούν από ορισμένα κράτη-μέλη. Εν πάση περιπτώσει, όλα τα κράτη-μέλη δεσμεύονται ως προς αυτούς τους στόχους. Και αυτό είναι ε, ένα στοιχείο ύψης της σημασίας για τη στρατηγική 2020. και αφορά και την τρέχουσα εργασία μας βεβαίως. Το θέμα του ανοιχτού συντονισμού μας απασχόλησε και μας απασχολεί. Ε, έχουν διαγραφεί αρκετές ανεπάρκειες. Θα πρέπει να βελτιωθεί αυτός ο ανοιχτός συντονισμός και θα ενταχθεί στις ε, μελλοντικές μας εργασίες. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα τη στιγμή που δεν έχουμε επιτάπητος μία στρατηγική. Ως προς την διαμεσολάβηση για τη φορολογική συνιστόσα, δηλαδή ποιες είναι οι φορολογικές απόρριες μίας απόφασης, θα μπορούσα να πω ότι σύμφωνα με το ΕΚΟΦΗΝ, εάν υπάρχει δεσμευτική απόφαση για μια Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή, αυτή η δεσμευτική απόφαση θα μπορούσε να αμφισβητηθεί από ένα κράτος μέλος εάν έχει φορολογικές συνέπειες. Και αυτό είναι απόλυτα λογικό. Εγώ βεβαίως δεν μπορώ να προδικάσω μία επερχόμενη συμφωνία μετά τις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει όμως να σας πω ότι η συμφωνία σε επίπεδο ΕΚΟΦΗΝ θίγει αυτό το ζήτημα και μιλά για μια διαδικαστική πορεία. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχουν, υπάρχει μια φορολογική συνιστόσα, φορολογικές συνέπειες ή κατά πόσο πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια επίγουσα ανάγκη αποκλειστικά. Τέλος, ως προς θέμα της απασχόλησης, εντάσσεται στη βασική αυτή στρατηγική, στη βιώσιμη αυτή στρατηγική 2020, διότι η χρηματοπιστωτική κρίση σε μεγάλη απώλεια θέσεων εργασίας με σοβαρότερη επίπτωση σε ορισμένα κράτη-μέλη και θα πρέπει να μας σε αυτή η βιώσιμη αναπτυξιακή στρατηγική και υποκοινωνικούς όρους και γι' αυτό η Ισπανική Προεδρία προτείνει ένα μεγάλο κοινωνικό σύμφωνο γύρω από την στρατηγική ανάπτυξη. Όπως ξέρετε, ο Υπουργός Οικονομίας μίλησε για ορισμένες γενικότερες κατευθυντήριες γραμμές της προάλλες για τα διαρθρωτικά ταμεία, που θα διέπουν τα διαρθρωτικά ταμεία. Θα πρέπει να ορίσουμε προτεραιότητες. Πρόκειται για κανόνες συνοχής που θα διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Thank you very much. Now by chance, rather... Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, συμβαίνει κατά τύχη να υπάρχουν τρεις ισπανόφωνοι ερωτητέ και ερωτήτριες. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να σας καλωσορίσω να, να καλωσορίσω την Ισπανική Προεδρία, το θάρρος σας και το ευρωπαϊστικό πνεύμα που σας διέπει. Όπως ξέρετε, τώρα βγαίνουμε από τις συμπληγάδες, ίσως βγαίνουμε, ίσως όχι, και ίσως βρεθούμε σε πιο ήσυχα νερά. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μελλοντική μας πορεία, η οικονομική μας πορεία. Η στρατηγική της ε, Λισαβόνας δεν είχε τα κατάλληλα μέσα για να φτάσει στους στόχους της. Και υπάρχουν 20 χώρες οι οποίες γνωρίζουν πολύ υψηλό έλλειμμα, δηλαδή κακή κατάσταση των δημοσίων οικονομικών. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε και την επίλυση του θέματος του δημοσίου χρέους και την απασχολησιμότητα. Τι μπορούν να κάνουν αυτά τα κράτη, πώς να αντιμετωπίσουν την κρίση πώς να αναζωογονήσουν την οικονομία τους και πώς να οδηγήσουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με βάση τη στρατηγική της Λισαβόνας και τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές. Ευχαριστώ. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου. Θα σας υποστηρίξουμε ως πολιτική ομάδα για να επιτύχετε μια καλύτερη ρύθμιση χωρίς την οποία δεν μπορεί να αναπτυχθεί η χρηματοπιστωτική αγορά. Η ιστορία των κρίσεων καταδεικνύει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάκαμψη χωρίς να εξηγιάνουμε την κατάσταση των τραπεζών. Ο Ντομινίκ Στρόσκαν, ο πρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τόνισε ότι δεν έχουν εξυγιανθεί οι τράπεζες. Και το πρόβλημα αυτό είναι περισσότερο ευρωπαϊκό παρά αμερικανικό. Τη στιγμή που εμείς ε, κατέχουμε, έχουμε τη θέση της Προεδρίας, πώς θεωρείτε μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Την προηγούμενη εβδομάδα η Τράπεζα της Ισπανίας δημοσίευσε τον ισολογισμό της, αλλά κανένας δεν σχολίασε τις καταθέσεις στην Ισπανία. Από τον Ιούνιο μέχρι τον Νοέμβριο είχαμε μία μείωση της τάξης του 4%, κάτι το οποίο είναι κάτι το πρωτόγρονο για τα δημόσια οικονομικά μας. Σήμερα το Ταμείο Παρακαταθήκων της Ισπανίας τόνισε ότι δεν μπορεί να πληρώσει το χρέος της και αυτό θα έχει επιπτώσεις στο rating που θα μας δοθεί. Δηλαδή μιλάμε για ένα 30% του ΑΕΠ μας. Πώς μπορείτε να σχολιάσετε αυτές τις δηλώσεις. Η Ευχαριστώ. Καλωσορίσατε κυρία Αντιπρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλες τις πληροφορίες που δώσατε. Νομίζω ότι καθίσατε σαφές το ενδιαφέρον μας για τη στρατηγική 2020 η οποία διαγράφεται τώρα. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτή τη στρατηγική μέσα στα πλαίσια της απασχολησιμότητας και του συνταξιδοτικού. <clears throat> Σα eh, Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω εντάχει σε ερωτήσεις αυτές. Ως προς τη στρατηγική 2020, προσπαθούμε να εξέλθουμε από μία οικονομική κρίση και γι' αυτό ακριβώς οφείλουμε να ορίσουμε μία στρατηγική. πολλές χώρες αντιμετωπίζουμε υπέρογκο δημοσιονομικό έλλειμμα. Και γι' αυτό θα πρέπει να προβούμε σε μεταρρυθμίσεις για να βελτιώσουμε τον ενδυνάμει αναπτυξιακό μας ρυθμό. Κάθε κράτος μέλος ακολουθεί ένα συγκεκριμένο οικονομικό μοντέλο με το οποίο μπήκε ή θα βγει και θα βγει από την κρίση. Υπάρχουν ορισμένες χώρες που θα πρέπει να προβούν σε αλλαγές ως προς τα οικονομικά πρότυπα που ακολουθούν. Θα πρέπει να δούμε την ανταγωνιστικότητα, την εσωτερική ζήτηση, τις εξαγωγές, την παραγωγικότητα. Εξαρτάται από το πού βρίσκεται ο καθένας. Νομίζω λοιπόν ότι οι μεταρρυθμίσεις θα γενικευτούν σε κάθε χώρα. Θα πρέπει όμως να προβάλλουμε έναν αναπτυξιακό ρυθμό και ένα ρυθμό ανάκαμψης για να φτάσουμε στην εκπλήρωση των ε, χρονικών στόχων του Συμφώνου Σταθερότητας όπως ε, χρονικά όρια τα οποία έχουν δοθεί σε κάθε κράτος μέλος χωριστά. Στον, προς τον κύριο Τρεμόσα, απαντώντας, δεν θα ήθελα να αναφερθώ στη, σε ισπανικά στοιχεία, ειδικά. Είναι γεγονός ότι η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ε, αναγνωρίζει ό τα στοιχεία ενεργητικού γνωρίζουν μία πτωτική πορεία στην Ευρώπη. Βεβαίως υπάρχει και ε, απόκληση απόψεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το γνωρίζετε. Πιο απεσιόδοξο είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υπάρχει δηλαδή διχογνωμία καταρχήν, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η αναγκαιότητα μιας αξιολόγησης των ε, στοιχείων ενεργητικού στους ισολογισμούς. Οι ισολογισμοί που θα πρέπει να ακολουθούν ε, κοινά κριτήρια. Αλλιώς έχουν οι ισολογισμοί στις ΗΠΑ και αλλιώς οι ισολογισμοί στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε κοινά ε, πρότυπα αξιολόγηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Αυτό ακριβώς θα προσπαθήσει να προωθήσει η Ισπανική Προεδρία για να προβούμε σε μία σύγκληση κριτηρίων και να μην υπάρχει αυτή η απόκληση αξιολόγησης όπως ίσχυσε μεταξύ Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και Διεθνούς Νομισματικού ναι. Ταμείου. Ως προς τα άλλα ερωτήματα θα ήθελα να σας πω ότι ως προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα βασικό ρόλο διαδραματίζουν οι εθνικές εποπτικές αρχές πρωτίστως. Προς κυρία Άλβαρες θα ήθελα να αναφέρω το εξής. Η στρατηγική 2020 θα προβάλλει μία βιώσιμη ανάπτυξη σε, ως προς το περιβαλλοντικό σκέλος, το οικονομικό και το ενεργειακό σκέλος. Θα λάβουμε υπόψη δηλαδή και τις τρεις αυτές συνιστώσεις υπό την εποπτεία του όπως είχε οριστεί υπό την, ε, αρχικά υπό την εποπτεία του Φελίπε Γκονσάλες. Εμείς θεωρούμε ότι το συνταξιοδοτικό είναι ένα θέμα ύψης της σημασίας το οποίο θα μας απασχολήσει μεσοπρόθεσμα. Okay. Um, I've still got five speakers left. The next three are... Uh, Πέντε είναι ομιλητές. And Pascal Canfin. So, Mr. Fio. Ο πρώτος. Κύριε Αντιπρόεδρε, θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ και σας εύχομαι κάθε επιτυχία για το υπόλοιπο της θητείας σας. Θα ήθελα να υποβάλω τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά το, τον ενδυνάμει αναπτυξιακό ρυθμό της οικονομίας. Τονίσατε τη σημασία της ενδυνάμει αυτής ανάκαμψης, αλλά όπως μας είπατε, 20 από τα 27 κράτη-μέλη βρίσκονται σε κατάσταση αντιμετώπισης υπέρογκου δημοσίου ελλείμματος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ε, υποβοηθά την αναπτυξιακή αυτή πορεία την ενδυνάμει αναπτυξιακή πορεία ή θα πρέπει να τροποποιηθεί ή θα πρέπει να παραμείνει ως έχει και να εφαρμοστεί με αυστηρότητα. Επίσης, στην εισήγησή σας τονίσατε το γεγονός ότι θα πρέπει να υποπτεύσουμε την κατάσταση της Ελλάδας. Θα ήθελα να ρωτήσω ότι το εξής, πέρα από την Ελλάδα υπάρχουν και άλλες οικονομίες που χρειάζονται ειδική παρέμβαση η ειδική προσοχή όπως ισχύει τώρα για την περίπτωση της Ελλάδας. Αν λάβουμε υπόψη και τα διάφορα ratings και τις διάφορες βαθμολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που έχουμε δει μέχρι ε, τούδε. Ως προς το φορολογικό καθεστώς, συζητήθηκε ο φόρος Τόμπιν πολύ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι γνώμη έχει το Συμβούλιο του, του θέματος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, και εγώ εξ ονόματος του ΕΛΚ του οποίου είμαι συντονιστής σας καλωσορίζω και εύχομαι η Ισπανική Προεδρία να αποφέρει αποτελέσματα. Εγώ δεν θα σας μιλήσω οικονομικά αλλά μεθοδολογικά, ίσως είναι γαλλικός τρόπος αυτός. Αν θέλετε να πετύχει η Προεδρία αυτή, θα έπρεπε να φέρει σε αποτέλεσμα τα, τις προθέσεις που έχει δηλωμένες. Αυτό σημαίνει να βρεθούν λύσεις από την πρώτη ανάγνωση. Ποιο, ποιος είναι αυτός ο τρόπος δεν είμαι παλαιός ευρωβουλευτής, αλλά ήμουν βουλευτής στη χώρα μου. Πρέπει να υπάρχουν πάντοτε κατάλληλα περιθώρια ελιγμών. Και τώρα που ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας, μην ξεχνάτε ποτέ ότι το Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτης. Και επομένως είμαστε καταδικασμένοι είτε να συνεννοούμαστε είτε να μπλοκάρουμε την πρόοδο της Ευρώπης από κοινού. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε όσο χρόνο χρειάζεται για μια σωστή διαπραγμάτευση για να βρεθούν ρεαλιστικές και πραγματιστικές λύσεις όχι μόνο για τα δημοσιονομικά αλλά και για το γενικότερο οικονομικό συμφέρον. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι σύντομο. Σε ποιο βαθμό είστε αποφασισμένοι να πετύχετε τις διαπραγματεύσεις με αυτό το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων που έχουν ίσες εξουσίες. Πασχάλης. Ευχαριστώ κυρία Υπουργέ. Επανέρχομαι στην ερώτηση των πρασίνων. Ίσως υπήρξε πρόβλημα μετάφρασης, αλλά δεν απαντήσατε ακριβώς. Ξέρω ότι έχετε διπλωματικούς κανόνες που πρέπει να εφαρμόσετε, αλλά υπάρχουν και οι δημοκρατικοί κανόνες που εφαρμόζουμε εμείς και που απαιτούν κάποια διαφάνεια. Για το θέμα των οικονομικών ανισοτήτων στην Ευρώπη και ανισορροπιών. Ως πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών θεωρείτε ότι τα ελλείμματα ορισμένων χωρών έχουν επιπτώσεις στο σύνολο των αποτελεσμάτων της Ευρωζώνης και ανατρέπουν το σύμφωνο σταθερότητας ή όχι. Και δεύτερον, αν σε μια χώρα η ιδιωτική χρέωση ας πούμε για τις αγορές ακινήτων έχει στρεβλώσει τα πράγματα. Θεωρείτε ότι τότε η πολιτική θέση του Συμβουλίου ως προς τον συστημικό κίνδυνο επιτρέπει τη δημιουργία σε αυτή τη χώρα μιας νέας έκρηξης όπως η παλαιότερη η προηγούμενη κρίση. Και τι θα κάνετε αν το Συμβούλιο δεν ανταποκριθεί έτσι. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Δεν είναι θέμα, δεν τίθεται θέμα διπλωματίας. απλώς συντονίζω δραστηριότητες του Συμβουλίου μέσα στα πλαίσια της εξαμηνίας Προεδρίας και προσπαθώ να τηρήσω τις κατευθυντηρίες γραμμές του Συμβουλίου. Σε σχέση με την ενδυνάμει αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας και το, τα υπέρογκα ελλείμματα, κατά πόσο δηλαδή το σύμφωνο σταθερότητας αρκεί ως μέσον αντιμετώπισης των υπέρογγων ελλημάτων και του δημόσιου χρέους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι προσετέθηκαν μία σειρά συστάσεων προς διάφορες χώρες με βάση το Σύμφωνο Σταθερότητας. Υπάρχει μία συνοδευτική σειρά συστάσεων προς τις χώρες με υψηλό έλλειμμα, έτσι ώστε να ανταποκριθούν μεσοπρόθεσμα, να αντιμετωπίσουν το έλλειμμα και το έλλειμμα και το χρέος τους. Θεωρούμε ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας αποτελεί στοιχείο κλειδί για την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη ανάκαμψη, συγγνώμη. Ως προς το θέμα της Ελλάδας που με ρωτήσατε, κατά πόσο δηλαδή θα μπορούσε να υπάρξει μία παρέμβαση τύπου Ελλάδας και σε άλλες χώρες, θα ήθελα να πω ότι στην ε, ε, Ελλάδα βασιστήκαμε στις στατιστικές. Η Eurostat βρέθηκε in situ όπου έγιναν ορισμένε επαληθεύσεις και μετά προβλήθηκε ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα υποβληθεί στο επόμενο ΕΚΟΦΗΝ για τη βελτίωση των στατιστικών στοιχείων. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει κανένας άλλος παρεμβατισμός ή παρέμβαση πέρα από τη διόρθωση των στατιστικών στοιχείων. Σε σχέση με την φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, το τέλος τόμπιν είναι μία πρόταση η οποία ε, προβλήθηκε και υπάρχει επιτάπητος και είναι μία πρόταση που απασχολεί όλα τα κράτη-μέλη. Θεωρούμε ότι θα ήταν αποτελεσματικό αυτό το μέτρο μόνο αν επιβαλόταν σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό πιστεύω ότι τα μέτρα που θα μας απασχολήσουν θα είναι μέτρα ευρωπαϊκής εμβέλειας και όχι εκτός ευρωπαϊκής εμβέλειας. Αυτό μέσα στα, πλέτη, πλαίσια ενός άτυπου συμβουλίου, διότι μιλάμε για την σχετική αποδοτικότητα του καθενός μέτρου χωριστά. Επαναλαμβάνω τα λόγια του Επιτρόπου Κόβαξ στο τέλος του ΕΚΟΦΗΝ ο οποίος είπε ότι εγώ δεν θα στοιχηματίζα ε, υπέρ ενός τέτοιου μέτρου, ότι θα μπορούσε δηλαδή να, να τύχει ε, θετικής αποδοχής και να οδηγεί σε ευημερία ένα τέτοιο μέτρο. Η εφαρμογή του είναι καθόλου εύκολη. Ως προς τα περιθώρια ελιγμού, Νομίζω ότι όσα μέσα έχουμε στη διάθεσή μας, όσα περιθώρια θα τα χρησιμοποιήσουμε, διότι η χρηματοπιστωτική κρίση και οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε μας οδηγούν στο να είμαστε πεπισμένοι ότι χρειάζεται μεγαλύτερη πεποπτεία. Εποπτεία η οποία θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή το ταχύτερο δυνατόν. Άρα θα ασχοληθούμε με την οδηγία που σας απασχόλησε και εσάς με μια έκθεση. Θα ασχοληθούμε με τις εποπτικές αρχές και εμείς έχουμε τη θέληση να φτάσουμε σε μια συμφωνία το ταχύτερο δυνατόν. Τέλος, ως προς τις ανισομέρειες, τα, τις ε, φούσκες, τις κερδοσκοπικές φούσκες, εμείς κινηθήκαμε στην Ευρωζώνη, στο Eurogroup, διότι υπάρχει θέμα σχετικής ανταγωνιστικότητας και υπάρχει και η σχετική τεκμηρίωση επί του θέματος. Έγινε λόγος για μεγαλύτερες ανισορροπίες και ανισομέρειες, λαμβάνοντας υπόψη και τις αναδιόμενες οικονομίες. Η λύση δεν έγκυται, δεν έγκυται σε εμάς. Μπορούμε να μιλήσουμε για μέτρα έτσι ώστε η Ευρώπη να είναι πιο ανταγωνιστική μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής 2020, αλλά οι λύσεις δεν είναι καθόλου εύκολες. Μιλήσατε για την ισπανική περίπτωση για την ε, πιστοληπτική ευκολία που υπήρχε στην Ισπανία και για τα επιτόκια που ήταν πολύ χαμηλά έως και αρνητικά και γι' αυτό δημιουργήθηκαν και αυτές ε, οι φούσκες στην κτηματαγορά. Αυτό έχει σχέση και με το γενικότερο πλαίσιο διαχείρισης της εγγύου ιδιοκτησίας. Δεν υπάρχει ένας ε, μόνο υπέτειος. Αυτές όμως οι φούσκες της κτηματαγοράς υπήρχαν και θα υπάρχουν και διέπουν αυτή την κρίση. η Αρλή Μακάρθη και μετά η Άννη Ξέρω ότι περιλαμβάνει η πολιτική σας και τα θέματα των αμοιβών των αποζημιώσεων. Έχουμε και το σχετικό κείμενο για τι ελάχιστε απαιτήσει για την οικονομική σταθερότητα. Ήθελα να ρωτήσω, υπό το φω τη ε, ε, συζήτηση που γίνεται για τα μπόνου και τι αποζημιώσει και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στι εξεχωριστέ ε, δράσει που έχουν αναλάβει τα κράτη-μέλη, θα συμφωνούσατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οδηγία της θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξη και θα πρέπει να βελτιώσει τις πολιτικές για τις αποζημιώσεις και η Ισπανική Προεδρία θα ξανασυζητήσει το θέμα αυτό των αποζημιώσεων στα πλαίσια της συζήτησης που γίνεται και σε συνεργασία με την σχετική Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και σας κυρία Αντιπρόεδρε για τις εισαγωγικές σας παρεμβάσεις και τοποθετήσεις. Ήθελα να μείνω λίγο στην υπόθεση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Αναφέρθηκαν πάρα πολλοί συνάδελφοι. Είναι γνωστό ότι πολλές χώρες, 20 και παραπάνω χώρες, αντιμετωπίζουν θέμα με τα δημόσια οικονομικά τους. Θέμα υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος είναι ένα μείζον θέμα για την Ευρώπη και ειδικά για την Ευρωζώνη. Αναφερθήκατε ωστόσο, κυρία Υπουργέ, ονομαστικά στην Ελλάδα και ασφαλώς δεν ήταν η πρώτη φορά. Ε, και μιλήσατε για το ενδεχόμενο απόσυρσης της ε, δημόσιας υποστήριξης εάν αποδόθηκαν ε, σωστά αυτά που είπατε και για μια νέα αρχιτεκτονική επιτήρησης που θα συζητηθεί στο επόμενο ΕΚΟΦΗΝ. ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν με δεδομένο ότι υποβλήθηκε πολύ πρόσφατα ένα τριετές επικαιροποιημένο πρόγραμμα σταθεροποίησης και ανάπτυξης από την νέα ελληνική κυβέρνηση που έτυχε κάποιας, ευνοική ευνοϊκής υποδοχής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και, από τον ε, προεδρεύοντα του, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και επειδή ε, αντιλαμβάνομαι ότι το θέμα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, είναι ευρύτερο, ε, ποια είναι τα επόμενα βήματα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι ε, ακριβές αυτό που είπατε πριν ότι υπάρχει θέμα απόσυρσης της δημόσιας υποστήριξης και υπό ποιες προϋποθέσεις. Το ένα ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα που θέλω να σας υποβάλω έχει να κάνει ε, με τα μεγάλα, τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες με υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα απέναντι στις αγορές, ότι είναι κατά κάποιο τρόπο εγκαταλελειμμένες στο έλεος των αγορών, ότι το κόστος του δανεισμού, το κόστος του χρήματος ανεβαίνει στα ύψη, γίνονται θύματα πολύ εκτεταμένων κερδοσκοπικών παιχνιδιών με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο η προσπάθεια για τον περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος. Επειδή αυτό θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που ε, το υφίσταται σήμερα η Ελλάδα, αλλά είναι ευρύτερο πολιτικό σοβαρό θέμα, ήθελα να σας ρωτήσω αν σας προβληματίζει ε, και αν θεωρείτε ότι χρήζει ε, κάποιας αντιμετώπισης. Σας ευχαριστώ. <clears throat> Σε σχέση με τις ε, πολιτικές αμοιβών, οι οποίες ε, δεν συμπεριλαμβάνονται στην ε, οδηγία κεφαλαιακής επάρκειας, το θέμα αυτό μας απασχόλησε στο Συμβούλιο. Ορίσαμε ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές και η πρόταση οδηγίας προβάλλει απαιτήσεις προς τους φορείς αυτούς για να βελτιστοποιήσουν τις πολιτικές αμοιβών και να μην τις αντιμετωπίζουμε μόνο βραχή πρόθεσμα. Γιατί η πολιτική υπερβολικών κινδύνων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και ακριβώς λέμε ότι θα πρέπει να ελέγξουμε και την πολιτική αμοιβών. Πολλές φορές με το θέμα ασχολούνται οι εθνικές εποπτικές αρχές. Γνωρίζετε την περίπτωση της Ισπανίας όπου οι εποπτικές αρχές της Κεντρικής Τράπεζας απασχολούνται και με τις πολιτικές, την πολιτική αμοιβών, ορίζουν την πολιτική αμοιβών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Εδώ υπάρχει μία πολιτική συστάσεων στην Ευρωπαϊκή Οδηγία. Ως προς το θέμα της Ελλάδας θα ήθελα να σας πω ότι ότι δεν θα αποσυρθεί καμία υποστήριξη, θα υπάρξει υποστήριξη και το λέω και το τονίζω. Και το μόνο στο οποίο αναφερθήκαμε ήταν τα στατιστικά στοιχεία. Βασιστήκαμε στα στατιστικά στοιχεία. Δεν υπάρχει καμία ε, άλλη επίπληξη ή παρεμβατισμός. Το θέμα είναι το δημόσιο έλλειμμα. Και το Φεβρουάριο θα ε, παρακολουθήσουμε την κατάσταση σε σχέση με το υπερβολικό έλλειμμα. Αλλά δεν υπήρξε καμία άλλη μορφή ε, δράσης ή επίπληξης. Θα υπάρξει μία σειρά συστάσεων, ως ήθιστε, και στα επόμενα συμβούλια του ΕΚΟΦΗΝ θα παρακολουθήσουμε την κατάσταση. Ακούσαμε βεβαίως και τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών και γνωρίζουμε ότι θα δοθεί συνέχεια. Στη συνέχεια η Επιτροπή θα συντάξει μία έκθεση για το επόμενο ΕΚΟΦΗΝ. Καμία άλλη δράση ή μορφή δράσης δεν προβλέπεται. Ούτε καν έγινε λόγος γι' αυτό τα συμπεράσματα του Συμβουλίου βασίζονται στα στατιστικά στοιχεία της Ελλάδας, αποκλειστικά και καθαρά. Και νομίζω ότι σας απάντησα. Τώρα, ως προς το κατά πόσο οι χώρες μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μείωσης του ελλείμματος, αυτό είναι ένα ζήτημα που θα το δει το χωριστά και θα πρέπει να τον λαμβάνει υπόψη τη στιγμή που προβάλλει ένα σχέδιο οικονομικής δραστηριότητας. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ε, πίασαμε αρκετά για θέματα που ε, μερικές φορές ε, την χάνουν κάποιων έτσι, μυστικών διαπραγματεύσεων. Μας είπατε εσείς κάποια πράγματα. Ελπίζω να μπορέσετε να ε, επανέλθετε στην Επιτροπή μας στις 16 Μαρτίου, όπου θα Έχουμε την ε, συζήτηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα ήταν μεγάλη μας τιμή να σας ε, ξαναέχουμε ε, εδώ στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις απαντήσεις που μας δώσατε. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου και βεβαίως θα παραστώ στις